Καλημέρα συνάδελφοι, πολύ χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι εδώ μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Και ο Ρωμαίο Φράνς, καλώς ήρθε που είναι νέος εδώ. Οπότε σας καλωσορίζω όλους. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Έχω διάφορε σύντομε ανακοινώσει πριν πούμε στην ουσία. Πρώτα απ' όλα έγκριση των πρακτικών. 27-28 ε, ε, Ιουλίου, Αυγούστου. Αν δεν υπαρχουν αντιρρησει αντιρρήσεις, 27-28 Νοεμβρίου του 17, 19 Οκτωβρίου του 17, 4 Σεπτεμβρίου του 17, 31 Αυγούστου του 17, 20 22 Ιουνίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσει μέχρι το τέλο θα εγκριθούν. Ε, δεν έχουμε κροατικά, δανέζικα, μαλτέζικα και γκέλικ. Ε, οι συστάσεις των συντονιστών επίσης ε, θα πρέπει να μας πείτε αν υπάρχει καμιά διαφωνία. Τώρα, έχουμε πρόταση κανονισμού για τις εξελίξεις στη γειτονία, το μέσο συνεργασίας. Εγκρίνεται τον ορισμό συγκίτρας της κυρίας Σπινέλη και μετά όσον αφορά της κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. 17 Ιουλίου του 2018 η Γραμματεία της ΛΥΜΠΕ κυκλοφόρησε τον κανονισμό της 13ης Ιουλίου σχετικά με τον κανονισμό 515 κάθετος του 2014 όσον αφορά επιπλέον χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου-εξόδου ενημερώθηκαν τα μέλη από τη Γραμματεία ότι θα υπάρξει κοινοποίηση ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και ότι επεκτείνεται η προθεσμία για δύο μήνες μέχρι τη 13η Νοεμβρίου 2018 για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ελέγξει την κατάσταση και θα ισχύσει για δύο μήνες η παράταση αυτή από τις 13 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Τώρα, η προθεσμία εσωτερική για κάποιο μέλος της ΛΥΜΠΕ που θέλει να υποβάλει κάποια ένσταση είναι η 30 Αυγούστου 2018, 12 το μεσημέρι. Αν θέλετε να υποβάλλετε ε, ένσταση, παρακαλώ με email στείλτε την ένστασή σας στον πρόεδρο και στη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ πριν λήξει η προθεσμία. Επίσης, τη 10 Αυγούστου του 2018 η γραμματεία Τη Λύπη Κυκλοφόρηση απόφαση του Συμβουλίου με επέκταση δύο μηνών της περίοδου ένστασης για το κατεξοδότηση κανονισμό 1042 κάθετος 14 της 25ης Ιουλίου σχετικά με τον κανονισμό 514 κάθετος 2014 για τον ορισμό και την διαχείριση των αρμοδιοτήτων ελέγχου των αρμοδίων αρχών όσον αφορά τις ε, υποχρεώσεις και το καθεστώς των ελεκτικών αρχών. Η νέα περίοδος ελέγχου είναι για δύο μήνες από τις 16 Ιουλίου του 2018. Τα έγγραφα αυτά τα πήρατε από την ε, ΛΥΜΠΕ το newsletter της δηλαδή 24 Αυγούστου 2014. Η προθεσμία λοιπόν είναι 27 Αυγούστου 2018 στο 12 το μεσημέρι. Τρίτον, 21 Αυγούστου 2018 η Επιτροπή ενέκρινε νέα κατεξοδότηση πράξη. Πρόκειται για τον κατεξοδότηση κανονισμό 2015-849 και 2016-1675 όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάνου στο κατάλογο του σημείου 1 του παραρτήματος. Θα έχετε πάρει τα έγγραφα αυτά στο newsletter μας πάλι στις 24 Αυγούστου. Επίσης, οι Λίμπη και οι ΕΚΟΝ έχουν ε, επιμερισμένη αρμοδιότητα για το φάκελο αυτό και εφαρμόζεται το άρθρο 55 του κανονισμού. Αν έχετε αντιρρήσεις, ενστάσεις κτλ. πρέπει να τις υποβάλλετε μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το τέλος των εργασιών εκείνη την ημέρα δηλαδή. Έπειτα διορθωτικό στην κατεξοδότηση πράξη. 28 Αυγούστου 2018 η Επιτροπή έστειλε διορθωτικό ε, όσον αφορά τον ε, κατεξουδότηση κανονισμό της Επιτροπής 1042 του 2014, της 25ης Ιουλίου του 2014, σχετικά με τον κανονισμό 514 κάθος 2014, όσον αφορά τον ορισμό και τη διαχείριση των αρμοδιοτήτων ελέγχου των αρμοδίων αρχών και όσον αφορά το καθεστώς και τις υποχρώσεις των ε, Ελεκτικών αρχών. Σύμφωνα με την επιστολή της συνοπτικής διαδικασίας, το διορθωτικό αυτό αφορά μη ουσιαστικά ασφάλματα στις γλωσσικές εκδόσεις των τσεχικών και των κρατικών. Τώρα, 9 Αυγούστου 2018, το Κοινοβούλιο πήρε σχέδιο ε, εφαρμοστικής ε, απόφαση της Κομισιόν για τα μέτρα όσον αφορά το κατάλογο των ατόμων ε, στο πλαίσιο του συστήματος εισόδων-εξόδων το, η βασική πράξη είναι ο κανονισμός 2017-2226 για την καταγραφή των δεδομένων εισόδου-εξόδου των υπηκών τρίτων χωρών που ε, περνούν τα σύνορα των χωρών μελών και καθορίζει τις ε, συνθήκες και την νομοθεσία που ισχύει και υπάρχει και τροποποίηση τη σύμβαση που εφαρμόζει τη Συμφωνία Σέγγεν και τον κανονισμό 767 κάθε 2018. Ανακοινώθηκε στα μέλη της ΛΥΜΠΕ μέσω του newsletter της 24ης Αυγούστου. Αν υπάρχουν ε, ενστάσεις, παρακαλώ στην γραμματεία της ΛΥΜΠΕ πριν τις 30 Αυγούστου του 2018 στο 12 μεσημέρι. Τέλος, θα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 9 και 20 σήμερα. Γι' αυτό παρακαλώ να έχετε μαζί τις κάρτες σας. Καλώς, αυτέ ήταν οι ανακοινώσει για σήμερα το πρωί. Καλώς ήρθατε. Αυτέ ήταν οι ανακοινώσει μου. Αρχίζουμε τώρα, μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές, με τα θέματα ουσία στην ημερήσια διάταξη. Καταρχήν, αποστολή τη Επιτροπή Λίμπε στη Βουλγαρία. Κοινή επιχείρηση του Frontex. Η αποστολή έλαβε χώρα 12 με 14 Φεβρουαρίου του 2018. Έχουμε την παρουσίαση από την κυρία Βερζιά, που ήταν επικεφαλή. Οπότε έχετε και το λόγο, κυρία Βερζιά, παρακαλώ. Κριστίν, θα μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πέντε λεπτά έχω στη διάθεσή μου, έτσι. Λοιπόν, πήγαμε στη Βουλγαρία για να δούμε πώς πάει η κοινή επιχείρηση με τις βουλγαρικές αρχές. Είναι κάτι συμβολικό για την εξέλιξη της εντολής της Frontex από το 2016 που ξεκίνησε στη Βουλγαρία ακριβώ. Ευχαριστώ λοιπόν την γραμματεία της Επιτροπής μας, την Κατρίνη Μπέρτ πάνω απ' όλα, για τη δουλειά της, για τις διευκολύνσεις που μας πρόσφερε παρά τις διάφορες αντιρρήσεις, τα κτλ. Ευχαριστώ πολύ και τους συμβούλους που συμμετείχανε, Βασέν, Μαρία, Κριστιαν και Παναγιώτα, που μας βοήθησαν πάρα πολύ και με πολύ εξυπνό τρόπο και πολύ αποτελεσματικά. Θέλαμε να επαληθεύσουμε κατά πόσο η συνεργασία αυτή πάει καλά ανάμεσα στη Frontex και τις βουλγαρικές αρχές. και θέλαμε να διαπιστώσουμε ότι τηρείται η νομοθεσία. Όχι μόνο αυστηρά ο έλεγχος στα σύνορα, θέλαμε δηλαδή να επαληθεύσουμε αν τα θεμελιώδη δικαιώματα τηρούνται. Και είναι σημαντικό, νομίζω ότι όλοι που πήγαμε εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος της Frontex είναι να διασφαλίσει και τα δύο, δηλαδή την τήρηση ολόκληρης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Στη Σόφια συναντηθήκαμε με την ε, Πρωτογιώτοβα που ήταν ε, πριν ε, συναδερφός μας, τον Υπουργό Εσωτερικών Ραντεύ. Συναντηθήκαμε με το σύνολο των βουλγαρικών αρχών κυρίως ε, με όσου ασχολούνται με τον έλεγχο των συνόρων, τα κέντρα της αστυνομίας για τον έλεγχο ανάμεσα Τουρκία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Συναντηθήκαμε και με τους υπεύθυνους από τη Frontex και όλους τους παράγοντες ε, τοπικούς και διεθνείς που ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Πήγαμε επίσης στο Καπτέντρεβο που είναι το διασυνοριακό πέρασμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγαμε μέχρι τα σύνορα δηλαδή στο τείχος ανάμεσα στην Τουρκία και τη Βουλγαρία, που ονομάζεται προσωρινός εξοπλισμός. Ξέρω ότι σε κάποιους αδέρφους αρέσει αυτή η ορολογία. Επιμένω λοιπόν σε αυτήν. Και επίσης, χάρη στην κατανόηση των βουλγαρικών αρχών, επισκεφτήκαμε και το κέντρο ξένο του Πετικέτ που δημιουργήθηκε το 2011 με ευρωπαϊκά χρήματα. Ήταν σημαντικό για μας δηλαδή να τα έχουμε δει όλα αυτά. Ευχαριστώ λοιπόν τις βουλγαρικές αρχές, όσους μας υποδέχτηκαν, γιατί πραγματικά μας υποδέχτηκαν πολύ καλά και είχαμε έναν πολύ καρποφόρο διάλογο μαζί τους. Ευχαριστώ επίσης και για την διαφοροποίηση που είχαμε όσον αφορά τους συνομιλητές μας. Ε, η ιεραρχία με πολύ ευκολία μας υποδέχτηκε, δέχτηκε να μιλήσει μαζί μας τόσο στα σύνορα όσο και στο κέντρο για τους ξένους στο Ubinet. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο απολογισμός είναι γενικά θετικός. Και ότι όλοι οι συνομιλητές μας μίλησαν για την πρόσθετη αξία που προσφέρει η συνεργασία με την Frontex. Πήραμε απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις μας παρόλο που παραμένουν ε, κάποιες γκρίζες ζώνες, κάποιες σκιές. Μερικές φορές είδαμε να αποφεύγουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας. Για όλους αυτούς που περνούν τα σύνορα και κινδυνεύουν να σταλούν πίσω στην Τουρκία, έχουμε εκθέσεις και τις συζητήσαμε αλλά δεν πήραμε επαρκείς απαντήσεις. Δεν διαπιστώσαμε παραβιάσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια επίσκεψη σύντομη που είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς επακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Αναρωτιόμαστε επίσης για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άτομα τα οποία φαίνεται να ε, μπλοκάρονται στα σύνορα και κρατώνται 24 ώρες για να επαληφθεί ταυτότητά τους, η κατάστασή τους κτλ. Και πώς είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν άσυλο και πόσοι το παίρνουν στη Βουλγαρία. Και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στα κέντρα κράτησης, δεν ξέρουμε πόσες ακριβώς είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται για επιστροφή των ατόμων αυτών. Παρακολουθούμε την κατάσταση με την εξέλιξη και στην Τουρκία. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται ε, όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία με τη... μεταξύ Βουλγαρίας δηλαδή και Τουρκίας. Πολλέ ανησυχίε εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2016 στο ψήφισμά του για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και μάθαμε ότι υπήρχε ιστορικά συνεργασία ανάμεσα στις τουρκικές και βουλγαρικές αρχές από τη δεκαετία του 60 και που δεν έχει εξελιχθεί παρά την αλλαγή καθεστώτων εκατέρωθεν των συνόρων. Συνεπώς, πρέπει να πω ότι έχουμε ανησυχίες για περιπτώσεις επιστροφών γιατί μας είπαν ότι όταν ε, ε, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν από την άλλη μεριά των συνόρων ομάδες ατόμων, οι βουλγαρικές ε, αρχές ενημέρωναν τις τουρκικές, τις νοριακές αρχές, οπότε έτσι ήταν αδύνατον κάποιοι Τούρκοι να φτάσουν να ζητήσουν άσυλο. Έχουμε λοιπόν, εκφράσουμε κάποιους φόβους για τους κινδύνους. Και είναι αδύναμη αυτή η λέξη, έτσι, τους κινδύνους για τους Τούρκους που προσπαθούν να φύγουν από την Τουρκία, αλλά τελικά καταλήγουν στα χέρια των τουρκικών αρχών. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε το θετικό ρόλο της Frontex. Εκφράζεται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη έτσι, αλλά και για τον ρόλο κατάρτισης της. Ίσως πρέπει να επιμείνουμε για την κατάρτιση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα διαπιστώσαμε ότι η Βουλγαρία κάνει πολλές προσπάθειες για να ελέγξει τα σύνορα. Ίσως να εκφράσουμε τη λύπη μας για αυτό που μας είπαν και διαπιστώσαμε που είχε να κάνει περισσότερο με την παράτυπη μετανάστευση παρά με το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος. Μπορεί να εκφράσει κανείς ανησυχίες όταν φτάνουν πολλοί τουρίστες γιατί έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα στα σύνορα. Και εξάλλου το έχω ήδη πει και επιμένω για την τήρηση των, και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να μην υπάρχουν επιστροφές ατόμων. Αλλά θέλω να επιμείνω ότι αυτά που είδαμε στην αποστολή αυτή δείχνουν ότι η Βουλγαρία σέβεται σε μεγάλο βαθμό τις αρχές που ζητούμε από όλες τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν στο σύστημα Σέγγεν. Και όπως το έχει κάνει και η Επιτροπή πολλές φορές, έτσι και εγώ θα έλεγα ότι έφτασε η στιγμή η Βουλγαρία να ενταχθεί στο σύστημα Σέγγεν. Και προσωπικά θα πρότεινα να υπάρξει και άλλη αποστολή της ΛΥΜΠΕ για τα θέματα τα μεταναστευτικά και του δικαιώματος στο άσυλο γιατί κάπως μείναμε απογοητευμένοι, αλλά βέβαια η αποστολή μας δεν ήταν επικεντρωμένη σε αυτό κυρίως, αλλά στον έλεγχο των συνόρων. Αυτά, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για όλη αυτή την ενημέρωση. Πολύ σύντομα σχόλια, εάν θέλει κάποιος συνάδελφος που συμμετείχε στην αποστολή, Ο κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξέρετε που να ψηφίσουμε. Αλλά έχει περάσει καιρό και πραγματικά αυτή η αποστολή μας άνοιξε τα μάτια. Ως πολιτικοί έχουμε ακούσει πολύ ξελίνη γλώσσα για να θολώσουν τα νερά σε σχέση με το τι συμβαίνει. Όμως η επίσκεψη στη Βουλγαρία μας έφερε σε ένα άλλο επίπεδο γνώση. Το κέντρο κράτηση ήταν υποτίθεται για την προσωρινή στέγαση αλλοδαπών και τελικά μόνο προσωρινό δεν ήταν το κέντρο αυτό. Είδαμε τι γίνεται με τα προβλήματα από την οδηγία των επιστροφών. Οι άνθρωποι ουσιαστικά φυλακίζονται χωρί να γνωρίζουν καν ποιο είναι το νομικό, του, νομικό τους καθεστώς. Και όχι μόνο τα πρόσωπα που φυλακίζονται έχουν πρόβλημα, η ίδια κυβέρνηση αντιμετωπίζει πρόβλημα. Διότι αν δεν γνωρίζουν επακριβώ ποιο είναι το νομικό του καθεστώ, τι πρόσβαση έχουν στα ένδικα μέσα, καταλήγουν να φυλακίζονται για 18 μήνες. Και αν ξεφύγουν και βρεθούν στο δρόμο, τους ξανασυλλαμβάνουν. Δεν είναι καλό λοιπόν ούτε για τους ίδιου τους ανθρώπους αυτούς, ούτε για τα θεσμικά όργανα. Επίσης, με τις επαναπροωθήσει προ την Τουρκία, εάν δούμε στην άλλη χώρα τι γίνεται με τα με, τη, με, τα χιλιόμετρα, με την απόσταση κοντά στα σύνορα και ειδοποιήσει κανείς ε, τους Τούρκους συνοριοφύλακες ότι ε, βλέπουμε κόσμο να έρχεται προς τα σύνορα, μπορεί να είναι απλώς Τούρκοι πολίτες που προσπαθούν να ξεφύγουν από το καθεστώς της χώρας και τελικά καταλήγουμε να τους επαναπροωθήσουμε. Επίσης, το άλλο φανταστικό είναι ο, χάρτης, ε, ο φράχτης. Ο φράχτης που αποτίθεται ότι είναι μια μηχανική διευκόλυνση της κατάστασης. Τίποτε το πραγματικό εκεί σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης επώδυνο ήταν ότι ανακαλύψαμε ότι η κοινωνία των πολιτών, η κοινή γνώμη μα λέει ότι εφόσον η Frontex συμμετέχει σε όλε αυτέ τι εργασίε, τα πράγματα πάνε μια χαρά όπω πρέπει βάσει των κανόνων. Αν όμω η Frontex φύγει, τα πράγματα δεν ε, είναι σωστά. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ ε, είναι ότι δεν μπορεί ποτέ απροσδόκητα να αναλάβει δράση η Frontex. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να την προσκαλέσουν. Άρα αυτός ο φράχτης δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί, αλλά και για την διενέργεια των ε, επιχειρήσεων με σωστό τρόπο. Ευχαριστούμε κυρία Σαρχεντίνη. Δεδομένου όμως ότι έχει περάσει η ώρα, θα έλεγα να εγκρίνουμε το σχέδιο. Να ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα μέλη τη ε, αποστολή, τον κύριο Ράντεβ, Σάτινα, Στέτινα και την κυρία Φαγιόν. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά και να προχωρήσουμε στις ψηφοφορίες αν είστε όλοι έτοιμοι. Επίσης ε, κάτι το που πρέπει να πούμε από την αρχή ότι το ρολόι εδώ στα αριστερά μου δεν πάει σωστά, οπότε θα ξεκινήσουμε σε ένα λεφτό. Συνάδελφοι, αν είστε όλοι έτοιμοι να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Είστε έτοιμοι. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Αν είστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Σημείο 5. Γνωμοδότηση Λίμπε για το Γενικό Προπολογισμό του 2019. Ξεκινάμε με τις σχετικές τροπολογίες, τροπολογίε. τροπολογίες. Εισηγητής μα ο κύριος Χρυσόγονο δεν βρίσκεται εδώ. Εκπροσωπείται από την κυρία Κούνεβα για το οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία υπαριθμών 1, εάν η στολή έτοιμη. Τροπολογία. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Επιμέρους τροπολογίες δύο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Οκτώ πρώτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1B. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρία. Οκτώ δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Άρχεται. Πέρα. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 κάθετος 25 άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 32. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα επιμέρους τροπολογία 17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 6. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Η 31 απορρίφθηκε. Με συγχωρείτε. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 36. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 37. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 38. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 40. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική, άρχεται αυτή. Πέρας, εγκρίνεται 35 προς 8. Καμία αποχή. Και τώρα πάμε στις δημοσιονομικές τροπολογίες. Λίμπε 57-23, άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 5-6-5-1. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-63, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 5662. Άρχεται. Πέρας. 5664. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 5665. 56-65. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-66. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-67. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-68. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5703 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 5719 άρχεται. 5719 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5700 άρχεται. Πέρας Εγκρίνεται. 57-15. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 56-52. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 57-05. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-89-56-97 ταυτόσημες. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτονται. 56-87 και 56-96 ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτονται. 5702 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτονται. 5670 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-88, 56-98. Ταυτόσιμες. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 56-55. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-86 άρχεται, πέρας. Απορρίπτεται. 57-24 άρχεται, πέρας. Απορρίπτεται. 57-25 άρχεται, Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 56-84. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-85. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57-22 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-91 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57-04 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5674. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5675. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5676. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 57-33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-90. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56-77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56-78 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 5679. 56-79 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-80 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. 56-81 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56-82 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57-29. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57-30. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 5683. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5650. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. Ε, όχι, συγγνώμη. Πάμε στην συμβαστική 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-95. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 57-26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-92. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 5701. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 56-56 και 5694 που ταυτίζονται. Ψηφίστε παρακαλώ, αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 6. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Αρασχητή ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 35 υπέρ, 4 κατά και 3 αποχές. Ωραία, συνάδελφοι, περνάμε τώρα στο σημείο 6, ψηφοφορία για την έκθεση Σκρίπεκ για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες. Διαδικαστικά το πλαίσιο θα αλλάξει από τον Νοέμβριο του 2018 όταν και θα τεθεί σε εφαρμογή το, η νέα ευρωπαϊκή ε, νομοθεσία. Από εκεί και πέρα οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες θα προστίθενται στα παραρτήματα μέσω κατεξοδότηση πράξεων. Θέλετε το λόγο κύριε Σιγητά. Ναι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Και μεγάλο κίνδυνο συνιστούν οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες που πλέον πολλούνται και μέσω του διαδικτύου. Είναι ένας κίνδυνος τον οποίο πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας γιατί μεταξύ αυτών ε, βρίσκονται και ουσίες με πολύ περίπλοκα ονόματα, ονόματα όπως είναι η πρόπυλο φεντανίλη, μεθοξία και τελοφεντανίλη. 90 νεκρούς είχαμε πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτές τις ουσίες. Και αποτελεί κίνδυνο για όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία, για τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, για την αστυνομία και γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να υπερψηφίσετε την έκθεσή μου και εδώ και στην Ολομέλεια. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε τις ψυχοτρόπες ουσίες αυτές να, να πατήσουν πόδι στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Λοιπόν, περνάμε κατευθείαν, λέει ο Πρόεδρο, στην τελική ψηφοφορία, καθώ δεν λάβαμε τροπολογίε. Με ονομαστική κλίση «Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. 41 υπέρ, 1 κατά, 1 αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία απόφαση για έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων όσον αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κόσοβο. Η είναι η κυρία Τάνια Φαγιόν και θα ψηφίσουμε επί του σχεδίου έκθεσης που έχει συντάξει. Έχουμε μαζί μας και, τον, και την, τον, την Υπουργό του Κωσυφοπηδίου για Ευρωπαϊκά Θέματα. Ε, το σχέδιο έκθεσης ε, είχε πρώτο ε, υποβληθεί το Σεπτέμβριο του 2016 αλλά η ψηφοφορία για την, για την απόφαση έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων δεν είχε εγκριθεί. Υπάρχει όμως πλέον η, ε, η κύρωση από πλευράς Κωσοφοπεδίου της Διεθνούς Συμφωνίας με διάφορους συγκριτικούς δέκτες. Ε, στις 18 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των ε, υπολοιπόμενων συγκριτικών δικτών για την απελευθέρωση των θεωρήσεων και τον σχετικό οδικό χάρτη για το Κόσο. Ε, υπάρχουν λοιπόν ε, υπάρχουν κάποιες, κάποιες συγκριτικοί δείκτες όπως είναι η φύλαξη των συνόρων και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της ε, διαφθοράς ε, και έχουν πλέον έχουν ικανοποιηθεί και αυτοί οι κανόνες. Κύριε Φαγιόν θέλετε το λόγο με απόλυτη ψηφοφορία πλειοψηφία πρέπει να γίνει η, να υπερψηφιστεί η ψηφοφορία αυτή. Ήταν μεγάλη η διάρκεια και η διαδικασία αυτή για το κοσυφοπαίδιο και φέραμε να καταλήξουμε στη σημερινή ψηφοφορία. Είναι σημαντικό το βήμα αυτό για το Κωσόβο. Ε, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ε, αποκλεισμένο το κοσυφοπαίδιο από τη διαδικασία απελευθέρωσης θεωρήσεων και πρέπει να σας διαβεβαίωσω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά πάρα πολύ ε, εκτενέστατο έργο στην, ε, στο Κωσυφοπέδιο προκειμένου να μπορέσουν να ε, ικανοποιήσουν τους συγκριτικούς δείκτες που είχαμε θέσει. Γι' αυτό και θα ήθελα πραγματικά να σας παρακινήσω να υπερψηφίσετε αυτή την έκθεση γιατί πραγματικά το αξίζουν οι πολίτες της χώρας αυτής να έχουν πρόσβαση ελεύθερη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Τάνια. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στη ψηφοφορία. Μία ενιαία ψηφοφορία θα γίνει. Άρχεται η ψηφοφορία. Uh, and the is now closed. 30 υπέρ, 10 κατά, 2 εποχές. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην εισηγήτρια.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 Ωραία. Περνάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Πρόκειται για γνωμοδότηση. Συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο Εμίλιαν Πάβελ, σωστά. Α, αλλά η Πίργκετ Σίπελ θα μιλήσει εκ μέρους του Εμίλιαν Πάβελ. Πρόκειται λοιπόν για εξέταση των τροπολογιών όσον αφορά τη γνωμοδότησή μας για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Οπότε εκ μέρους του κύριου Πάβελ για πες μας Μπέργκετ τι λέει για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ Κλοντ. Ο Εμίλιαν δυστυχώς δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα, όπως είπες και εσύ, οπότε θα σας διαβάσω το σημείο που μου άφησε. Πρώτον, ευχαριστώ την Επιτροπή για την πρότασή της όσον αφορά τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Ευχαριστώ και την Επιτροπή Απασχόλησης. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική και από την πλευρά της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και αυτό αντικατοπτρίζουν οι τροπολογίες μου. Θα πρέπει να συνεισφέρουμε σε ενίσχυση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την διασυνοριακή κινητικότητα στα εργασιακά και να προστατευτούν και τα θεμελιώδη δικαιώματα βάσει των ε, κανόνων που μιλούν για την ε, διακίνηση, την ελεύθερη κυκλοφορία μάλλον των ατόμων μεταξύ των χωρών μελών. Στηρίζουμε επίσης την άσκηση των δικαιωμάτων και διασυνοριακά με σωστές και δίκαιες συνθήκες εργασίας, με ασφάλιση, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης ε, ανθρώπων. Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό της αδήλωτης εργασίας. Γι' αυτό και ο συγητής προτείνει τροπολογία που λέει πώς να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία που συχνά εμφανίζεται διασυνοριακά. Κάποιες πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι πήκοοι τρίτων χωρών, εκτίθενται ιδιαίτερα στην αδήλωτη αυτή εργασία και τους αρνούνται τα βασικά τους εργασιακά δικαιώματα. Γι' αυτό θα έπρεπε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις βάσω της πλατφόρμα μας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και να ενισχύσουμε περισσότερο την συνεργασία για τα εργασιακά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την προστασία δεδομένων, όσον αφορά την οδηγία 6791, και την 27 του 2001 που αναφέρεται στην προστασία δεδομένων, πρέπει να εφαρμόζονται στην ε, διαδικασία δεδομένων και με την πρόταση αυτή. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων περιορίζεται αναλογικά και βάσει ανάγκης και πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια νόμιμη ανάγκη και όχι να γίνεται με τρόπο ασύμβατο με τους κανόνες και πρέπει να είναι σαφές ότι οι αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει από κοινού να ελέγχουν τα θέματα της μεταφοράς δεδομένων. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η καταπολέμηση της απάτης. Εδώ πρόκειται για την εφαρμογή του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ανάμιξη του επόπτη δεδομένων όπου αυτό χρειάζεται εφόσον γίνονται έρευνες για παράνομη μεταφορά δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε, Μπίρκιτ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Είναι πολύ βασικά αυτά. Κανένας άλλος. Παρακαλώ, Τζιν Λάμπερτς. Ευχαριστώ πολύ. και ευχαριστώ για την παρέμβαση αυτή που κάνατε εκ μέρους του συντάκτη. Με τις τροπολογίες μας εμείς προσπαθούμε να περιοριστούμε περισσότερο στο ρόλο της ΛΥΜΠΕ, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως. Γιατί κυρίως η Επιτροπή Απασχόληση βέβαια είναι αρμόδια. Είμαι μέλος εκεί, αλλά δεν είμαι σκιώδης εκεί. Λοιπόν, και εμείς κοιτάξαμε τα θέματα αυτά που αναφέρθηκαν μόλις. Η διαδικασία επεξεργασία δεδομένων, για παράδειγμα, είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Και αυτό να το κάνουν οι υποπτικές αρχές πάνω απ' όλα, τον έλεγχο. Επίσης, το θέμα του Διαχειριστικού Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, θα έπρεπε να έχουν λόγο εδώ και πρέπει να αναφέρουμε και εμείς τι πιστεύουμε για το ρόλο τους, που είναι η ενίσχυση της κυκλοφορίας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Θέλουμε λοιπόν η κυκλοφορία αυτή να λειτουργήσει καλύτερα. Αλλά προσοχή, μην καταλήξουμε στο τέλος με μία αρχή που δεν έχει αρχή. Αλλιώς πρέπει να την ονομάσουμε αλλιώς, αν δεν έχει εξουσία. Να ξέρουμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει, ε, πώς θα γίνεται η διασυνοριακή συνεργασία, η επιθεώρηση και πώς θα λαμβάνεται δράση κάθε φορά που εντοπίζονται παραβιάσεις. Όποιος μπορεί να φέρει πληροφορίες θα πρέπει να μπορεί να το κάνει. Ε, εδώ όμως προσοχή δεν μιλάμε για μετανάστευση, μιλάμε μόνο για εργασιακά δικαιώματα, έτσι. Ναι, σωστά. Η κυρία Στίβενς. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για το έργο του. Συμφωνώ ότι πρέπει να σκεφτούμε καλά πώς θα προστατεύσουμε τα δεδομένα των ανθρώπων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για τους κινδύνους από το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τι γίνεται με την ανταλλαγή δεδομένων, ας πούμε των ε, κοινωνικών ασφαλίσεων. Επίσης, σωστά λέει ο εισηγητής ότι η συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρέπει να κάνει τέτοια πρόταση, όπως έγινε με τη Frontex. Αυτό που δεν μπορώ να στηρίξω είναι ότι μια τέτοια αρχή πρέπει να παρεμβαίνει και για θέματα που δεν είναι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν το θέλω καθόλου. πρέπει να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες δομές πρώτα απ' όλα πριν δημιουργήσουμε μια νέα αρχή. Αν όμως καταλήξουμε να έχουμε αυτήν τη νέα αρχή, θα πρέπει να προσφέρει μια προστιθέμενη αξία, γιατί στο κάτω-κάτω χρήματα θα κοστίσει. Και αυτή η πρόσθετη αξία δεν θα πρέπει να αφαιρεί κυριαρχία από τις χώρες μέλη. Και τέλος, πρέπει να σεβόμαστε τις αρμοδιότητες των χωρών μελών. Επιμένω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει προσθέμενη αξία από αυτήν την αρχή και να φροντίσουμε όντω να γίνονται κοινωνικές ε, έρευνες στα εργασιακά. Ευχαριστούμε κυρία Στίβεν. Στην τελευταία φορά που το συζητήσαμε αυτό το θέμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να πει την άποψή της. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάποιον. Ναι. Ωραία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και όλους τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο με συστάσεις και σχόλια ξέροντας ότι είμαστε αμέσω μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Όσον αφορά τις τροπολογίες, δεν θα μπω στην ουσία. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω ότι πίκο οι τρίτων χωρών περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή εφόσον καλύπτονται από την ομοθεσία κυκλοφορίας ασφάλιση κλπ. Στόχος της αρχής αυτής θα είναι να καταστήσει πιο αποτελεσματικούς τους οργανισμούς που ήδη υπάρχουν, είτε με συνεργασία, είτε με ε, βοήθεια την ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της αδήλωτης εργασίας θέλουμε να την ενσωματώσουμε εδώ προκειμένου και αυτή να λειτουργήσει καλύτερα να έχει στη διάθεσή της περισσότερα μέσα από όσα έχει τώρα. Όσον αφορά τώρα τον ε, στόχο των, της αρχής αυτής, φυσικά και πρέπει να είναι αποτελεσματική και αυτός είναι και ο στόχος μας, να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική αρχή που θα φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων, που θα βοηθάει τους εργαζόμενους, θα τους προστατεύει αλλά συγχρόνως καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλές αρμοδιότητες και κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα σχεδιάζονται έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη αυτή η ισορροπία. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και προσβλέπουμε σε παρετέρω συνεργασία μαζί σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μπίρκιτ, να προσθέσει κάτι, συμπέρασμα. Εννοείται ότι δεν μπορώ να πω τίποτα τώρα εκ μέρους του εισηγητή εγώ, όμως συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποια είναι τα καθήκοντα της νέας αυτής αρχής. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν, αν πρόκειται για συντονισμό, ας πούμε, όπως για την αδήλωτη εργασία διασυνοριακά, αλλά να είμαι σαφής. Πρέπει να γίνει πολύ περισσότερη δουλειά από πλευρά των χωρών μελών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, πρώτα απ' όλα. Οπότε, ναι, θέλω να περιγράψουμε τους στόχους και τις ε, αρχές της, ε, του νέου αυτού οργανισμού, προκειμένου να βοηθήσει να πάνε τα πράγματα καλύτερα από ό,τι πάνε τώρα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Καταλαβαίνουμε έτσι η ψηφοφορία θα είναι 10 Οκτωβρίου, σωστά. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας εδώ. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 9. Πρόκειται για τη μελέτη σχετικά με το κόστος της απουσίας Ευρώπης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα διακόψουμε όμως λίγο γιατί δεν έχουμε ακόμα εδώ τον αρμόδιο. Για λίγο έτσι. Μέχρι να έρθει εδώ. Ένα-δύο λεπτά, έτσι διάλειμμα. Uh, Συνάδελφοι, θέλω να δω και εσείς τι μου λέτε, να δω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα με το σημείο αυτό. Βρίσκονται εδώ οι δικοί μα. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, οπότε αν συμφωνείτε να ξεκινήσουμε, ωραία. Συνάδελφοι, μιλάμε για ακόμη σημαντική και ε, γεμάτη νόημα έκθεση, μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας και άπτωτα των αρμοδιοτήτων της. Και νομίζω το ζήτημα εδώ είναι εάν το υλικό που μας διδίθεται το αξιοποιούμε Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκπόνησή του και είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη και κέρια η έκθεση και η μελέτη για το κόστος της απουσίας της Ευρώπης στην καταπολέμηση της θερμοκρατίας. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την παρουσίαση αυτού ακριβώς ε, αυτής της μελέτης για, από την ερευνητική υπηρεσία, από την υπηρεσία ερευνών το κόστος της απουσίας της Ευρώπης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δηλαδή το τι γίνεται, το τι όταν δεν αναλαμβάνεται δράση σε πολιτικό επίπεδο. Κόστος ως προς τις υλικές φθορές και ζημιές. Η γραμμή που διατρέχει όλη την έκθεση είναι ότι υποτιμάται το κόστος αυτών των φθορών. Έχουμε εδώ λοιπόν δύο από τους συμπρογνωμονές μας τον έναν τον γνωρίζουμε καλά. Τον άλλον χαίρομαι που τον έχουμε ξανά. Τον κύριο Βούτερ, τον δόκτωρα μάλλον Βούτερ Φαν Μπάλεγκόι. Και τον δόκτωρα Χάφνερ από τη Rand Europe. Θα μας παρουσιάσουν την έκθεση. μια από τις μελέτες της υπηρεσίας ερευνών που μπορούμε να ε, αξιοποιήσουμε. Είναι ε, ένας αξιόλογος πόρος οι μελέτες αυτές και πρόκειται για ένα υλικό που μας είναι πολύτιμο για τη δουλειά της Επιτροπής μας. Βούτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πώ να αξιοποιήσετε τις εκθέσεις αυτές. Νομίζω το βασικό μήνυμα που προκύπτει είναι το κόστος της μη αναληψη δράσης. Όταν λοιπόν τα κράτη-μέλη περνάνε σε επιπλανατεύσεις και λένε αυτό κοστίζει πολύ αν εγκρίνουμε το τάδε το άλλο μέτρο, μπορεί κανείς να ε, προβάλλει αριθμούς και αριθμητικά στοιχεία για το κόστος, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά της μη ανάληψης δράσης. Ας πούμε, η ανισότητα, η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει οριζόντια οδηγία έχει κόστος στην καθημερινότητα των πολιτών και οικονομικό αντίκτυπο. Να ξεκινήσω λοιπόν με την παρουσίαση αυτή, όπως προσπαθήσω να τα πω ξεκάθαρα πριν μπω στην παρουσίαση της μελέτης αυτής, μια μελέτη που ενδιαφέρει πολύ ε, την δουλειά της Επιτροπής σας και για το χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ε, δικαίου που ζητήσατε από το 2016. Να πω ότι για μας που συνεργαζόμαστε με τους ομολόγους μας στην Washington όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έξι εκθέσεις που θα ε, ε, εκπονήσουμε και θα, τις, θα σας παραπέμψω σε αυτές γιατί θα τις αναφέρω καθώς τα συζητούμε εδώ. Τα δικαιώματα κατά την κράτηση, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και αυτό για το σύστημα ασύλου και των ελεγχών σύνορων, αλλά και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όλες αυτές οι εκθέσεις ακολουθούν τρία στάδια. Πρώτον, επισκόπηση της ε, υπάρχουσας κατάστασης και των νομικών ε, προβλημάτων και φραγμών στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον ε, εν λόγω χώρο κάθε φορά. Καινοτομία της έρευνας αυτής τώρα είναι ότι αποτιμάμε και τον οικονομικό αντίκτυπο του status quo. Οικονομικό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο Ως προ την κράτηση ας πούμε, των προσώπων, τι θεμελιώδει ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά παρουσιάζουμε διαφορετικές επιλογές για πολιτική δράση και το πώ θα μπορούσαν να αρθούν οι φραγμοί και να καλυφθούν τα κενά. Όλα αυτά ε, με την μελέτη που έχουμε και εσωτερικός αλλά και εξωτερικός. Σήμερα θα μιλήσω για τα κενά και τους φραγμούς στην καταπολέμηση της δημοκρατίας και τις διαφορετικές πολιτικές επιλογές και τα περισσότερα ε, στοιχεία θα τα δώσω ο κ. Χάφνερ. Από το Ευρωβαρόμετρο βλέπουμε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας παραμένει βασική μερίμνα των Ευρωπαίων πολιτών. Το αναφέρει 40% περίπου όσων ερωτηθήκαν το 2017. Παρόλο που βλέπουμε να υπάρχει μείωση πρόσφατα Κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ε, αντίληψη του κόσμου για το ότι είναι πρώτο θέμα προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η προστεθέμενη αξία τη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο και στι ευρωεκλογέ του χρόνου. Βεβαίω, Μιλούμε για αρμοδιότητε τη Επιτροπή Λίμπε σήμερα. Οπότε θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στο τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και στα πλαίσια των δικών σα αρμοδιοτήτων, κυρίω ε, από την ε, προσέγγιση τη ε, ελευθερία και δικαιοσύνη. Μικτέ αρμοδιότητε λοιπόν με τι κυβερνήσει των κρατών μελών. Πρέπει τα δύο επίπεδα, το ευρωπαϊκό και το εθνικό, να συνεργαστούν στενά. Πρέπει να υποστηρίξουμε εθνικά μέτρα και τι ανταλλαγέ μεταξύ των δύο. Πρώτα απ' όλα για την καταπολέμηση τη, την πρόληψη τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση. Μετά για την χρηματοδότηση τη ε, τρομοκρατία, τα όπλα και τα εκρηκτικά ε, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα τα δούμε και στην επόμενη έκθεση που θα εκπονηθεί από εμά. Έπειτα, ε, επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των, Ευρωπα... εθνικών διοκτικών αρχών, καθώ την εναρμόνιση τη ε, δράση για το για την δράση της Europol και όλων των σχετικών οργάνων, διοικητικών αρχών. Το ίδιο και στο ποινικό δίκαιο και την σχετική δικονομία πρέπει να υπάρξει περισσότερη εναρμόνιση καθώς και ενεργή συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο, υπάρχει και μια σειρά από κενά και φραγμούς που μπορούμε να εντοπίσουμε στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα ε, τα αποδεικτικά στοιχεία, η λογοδοσία και η επισκόπηση του πώς ε, σχεδιάζονται οι νόμοι και η αστυνομική συνεργασία στον τομέα αυτό. Ας πούμε πρέπει να γίνει υποσύνδεση μεταξύ της ε, επικέντρωσης στον, στην δημοκρατία των τζιχαντιστών, που είναι σχεδόν αποκλειστική, και μετά τις σημαντικές απειλές που προκύπτουν και από τους, ε, τις αποσχιστικές τάσεις τις ακροδεξιές και ακροαριστερές δημοκρατικές τάσεις, όπως δείχνουν οι εκθέσεις της Europol. Μεταξύ του 2001 και 2013, μεταξύ των 88 μέτρων κατά της τρομοκρατίας, μόνο ένα τέταρτο ε, ε, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτη αντικτύπου και μόνο τρία δημοσίων διαβουλεύσεων. Ακόμη και αν η κατάσταση έχει βελτιωθεί έκτοτε, και πάλι ε, μας έχει μείνει αυτή η παράδοση. Ως τώρα δεν υπάρχει σφαιρική ε, αξιολόγηση των μέτρων κατά της τρομοκρατίας. Ιδίως ως προς το κατά πόσον είναι εύστοχα, συνεπτικά, ε, αποτελεσματικά και ε, συμμορφούμενα με τις νομικές απαιτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπώνησε σφαιρική αποτίμηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, κάτι όμως διαφορετικό και είναι απλώς ένα θετικό πρωτοβήμα όλο αυτό. Επιπλέον, καταλήγουμε ότι οι μηχανισμοί επισκόπησης και παρακολούθησης της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην καταπολέμηση τη Δημοκρατία. Το δικαίωμα του Ευρωκοινοβουλίου να θέτει ερωτήσεις δεν μπορεί να ασκηθεί πλήρως ε, λόγω των εθνικών μέτρων και διαδικασιών, όπως με τα διάφορα εντάλματα που μπορεί να εκδοθούν σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά τα ερωτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως για την κράτηση και την, ε, τα φασανιστήρια σε υπόπτους για τρομοκρατία, αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω ερευνών και υπάρχουν και παραδόσεις ή ε, εκδόσεις που οδήγησαν και σε περαιτέρω εκδίκαση των υποθέσεων και σε, άλλα, σε άλλες δικαιοδοσίες και φόρα. Επίση, για τα προγράμματα ριζοσπαστικοποίηση και στατολόγηση. Τα πορίσματα μα δείχνουν ότι παρά την χρηματοδότηση τη έρευνα, ξέρουμε ακόμα πολύ λίγα για τα πραγματικά αίτια τη διαδικασία και του μηχανισμού που οδηγούν σε ριζοσπαστικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει σημαντικό ρόλο στην διάδοση των βέλτιστων πρακτικών, όμω η δράση αυτή ακόμα δεν συνοδεύεται από του απαραίτητου μηχανισμού παρακολούθηση με σωστή μεθοδολογία για να δούμε ποια είναι τα εθνικά προγράμματα, αν είναι αποτελεσματικά και αν συμμορφούνται με τι απαιτήσει για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η έκθεση δίνει και παραδείγματα για το πώ οι δημόσιε συζητήσει και οι πολιτικέ αντιμετωπίζουν το φαινόμενο ε, των ανθρώπων που αρχίζουν να ενστερνίζονται ιδεολογίε και απόψει, ή δόγματα που οδηγούν στην ριζοσπαστικοποίηση πολλέ φορέ σε σχέση και με θρησκευτικέ ε, απόψει Τέτοιε τοποθετήσει και εκφράσει δημιουργούν προβλήματα και κυρίω σε μέρη των, ε, του πληθυσμού που αποτελούν ήδη αντικείμενο μίσου και διακρίσεων. Σε σχέση με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων είδαμε τέσσερις περιπτώσεις ε, μουσουλμάνων ε, που αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης και μίσους αυτό το είχαμε συζητήσει και στην ε, περσινή μα έκθεση για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβία και είδαμε και το σχετικό κόστο που προκύπτει. Τρίτον, στον ε, χώρο τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, Εδώ πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των ε, καθηκόντων υποβολή εκθέσεων στον ιδιωτικό τομέα, τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών διώξεω οικονομικού εγκλήματο, με τι σχετικέ εκθέσει ανάλυση και τι διαδικασίε μεταφοράς ποσών βάσει και του σχετικού προγράμματος ταχείας ανείχνευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά δείχνουν ότι το πλαίσιο δεν είναι πλήρε. Ιδίω για τις ενδευρωπαϊκέ πληρωμέ σε ευρώ, καθώς για τις περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις δεν χρειάζονται μεγάλα χρηματικά ποσά τελικά. Επίσης το θέμα είναι και η συνολική συμμόρφωση με τις απαιτήσει για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η έκθεση ε, εντοπίζει ότι η συνεργασία των διοικητικών αρχών μέσω των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων δεν έχει φτάσει στο πλήρες δυναμικό της. Ξέρω ότι η Επιτροπή σας εργάζεται για το σκοπό αυτό. Είναι περίπλοκο το αρχιτεκτόνημα των βάσεων δεδομένων. Ε, λείπει η απαραίτητη διασύνδεση. Υπάρχουν νομικέ και τεχνικέ δυσκολίε. Αλλά λείπει και η προθυμία κάποιων εθνικών αρχών να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίε. Η έκθεση εντοπίζει ότι η αποτελεσματική δικαστική συνεργασία, όπω με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, τι κοινέ ομάδε έρευνα, υπονομεύεται από την έλλειψη συμμόρφωση με τι απαιτήσει των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπω α πούμε με τι ε, συνθήκε κράτηση. Αλλά δεν υπάρχουν και κοινέ ε, κοινοί ποινικοί ορισμοί για τα ένδικα μέσα ή τα εχέγγυα ή την προστασία των υπόπτων. Η Συνεργασία μεταξύ των ε, οργάνων των ε, εθνικών κρατών δεν είναι ακόμα πλήρως ε, οργανωμένη. Η αδερφότητα των δυνάμεων δράσης, ας πούμε, η φρατερνητέ όπως οργανώθηκε μετά τις επιθέσεις της Βρυξέλλες, είναι απλώς κάτι το άτυπο. Τώρα, στην επόμενη διαφάνεια λέω ότι πρέπει να δούμε ε, αυτά που ξέρουμε με βεβαιότητα, αυτά που δουλεύουν και αυτά που δεν δουλεύουν για την καταπολέμηση της δημοκρατίας. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα κύκλο κατάρτισης πολιτικής ευρωκοπέδου που να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία με τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν είναι καινούργια πρόταση αυτή. Ήδη Το είδαμε στην έκθεση με θέμα την απουσία της Ευρώπης στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Εάν λοιπόν δούμε την συνεργασία της δικής σας επιτροπής με τις άλλες αρμόδιες επιτροπές που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερη συνεργασία. Σημαντικό είναι ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει κάνει σχετικές προτάσεις για έναν πολιτικό κύκλο για την παρακολούθηση ε, του τι γίνεται στο κράτος δικαίου των θεμελιωτών δικαιωμάτων και του χώρου δικαιοσύνη. Γενικώ, και αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει στα πλαίσια του οργανωμένου εγκλήματο και τη διαφθορά, ένα κράτο μέλο που δεν αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά, διαφθορά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και την τρομοκρατία εύκολα. Οι κοινέ προσπάθειε θα πρέπει να γίνονται από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να καταλήξουμε σε μια σφαιρική αξιολόγηση των μέτρων καταπολέμηση τη τρομοκρατία με μελέτε αντικτύπου και αξιολογήσει και αποτιμήσει. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο παρακολουθώντα τι αποφάσει τη Επιτροπή για τη μη εκπόνηση μελέτη αντικτύπου. Η συνεργασία και τα εργαλεία που διατίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφύγουμε τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση στη τρομοκρατία και η έλλειψη συνεργασία πρέπει να μελετηθούν και να ενισχυθούν. Αυτό μπορεί να γίνει με την ανάπτυξη ενό σφαιρικού πολιτικού πλαισίου. Ξέρω ότι υπάρχουν σχετικέ προτάσει, ήδη, αλλά μπορεί να υπάρξουν και μηχανισμοί για την προκλήθηση των δράσεων των 100 μελών με βάση ξεκάθαρες μεθοδολογίες. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει το τι γίνεται ταυτόχρονα με τις εκπαιδευτικές πολιτικές, τις οικονομικές πολιτικές, τις κοινωνικές. Όπως είπαμε για τις συνθήκες κράτησης, πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης, να υπάρχουν περισσότεροι ε, υπάλληλοι αστυνομικοί που να ασχολούνται με τις ε, αναστολές, με την ε, παρακολούθηση της κράτησης πρέπει να τα δούμε και από τη σκοπιά, τη δικαστική και την ποινική. Εάν όχι, οδηγούμε και εμείς τους φυλακισμένους σε ριζοπαστικοποίηση. τελευταία διαφάνεια. Χωρίς χρηματοδότηση τρομοκράτες και μπορούμε να βελτιώσουμε το σχετικό πλαίσιο, και με την ενίσχυση των διοικητικών αρχών στα δεδομένα μπορούμε να βελτιώσουμε το συνολικό πλαίσιο. Το ίδιο και αν Το ίδιο και αν υπάρξει ένα σύστημα ανείχνευση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμω η δημιουργία ενό τέτοιου συστήματο μπορεί να γίνει στο επίπεδο τη ενίσχυση τη συνεργασία των διοκτικών αρχών. Και βεβαίω πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ομολογία του ΔΕΚ. Τέταρτον, πρέπει να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα συνεργασία των διοκτικών αρχών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι, πιο κέρδε πληροφορίε να είναι αυτέ που ανταλλάσσονται υποστηρίζοντας τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό για να γίνεται με ε, τρόπο φυσικό. Όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα μακροπρόθεσμο. Δεν μπορούμε μόνο με τεχνικά μέτρα και συνδρομή, αλλά χρειάζεται και περαιτέρω χρηματοδότηση για να γίνουν όλα αυτά. Τώρα είναι η τελική διαφάνεια για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την τρομοκρατία. Τα μέτρα που έχουμε προτείνει θα πρέπει να βελτιώνουν την ε, καλή ε, διαβίωση του πληθυσμού, να αντιμετωπίζουν πραγματικά την τρομοκρατία και να έχουν και κάποιο αντίκτυπο στην πραγματικότητα. Περισσότερε λεπτομέρειε θα σα δώσω συνάδελφο σε ένα λεπτό. Για περισσότερε λεπτομέρειε μπορείτε να πάτε και στον σύνδεσμο που περιέχεται στην έκθεση. Um, Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ραντ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία σήμερα να σας μιλήσω για το κόστος ε, της τρομοκρατίας και των ε, σχετικών ε, αντιτρομοκρατικών μέτρων που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί σε τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Ακόμη περισσότεροι άνθρωποι όμως ε, επηρεάζονται και πλήττονται ε, από τέτοιου είδους τρομοκρατικές ε, επιθέσεις πέραν των άμεσων θυμάτων. Και αυτό είναι και ο βασικός στόχος τρομοκρατίας, η διάδοση του φόβου. Να διαταραχθεί δηλαδή, να διαταραχθούν οι θεσμικές, δημοκρατικές, πολιτικές δομές μιας κοινωνίας. Και έτσι υπάρχει μια πλειάδα επιπτώσεων στους πολίτες. Σκεφτείτε όλα τα μέτρα ασφαλείας, σε αεροδρόμια, σε κυβερνητικά κτίρια, τους συνοριακούς ελέγχους που μπορούν επίσης να επλήξουν την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα. Γι' αυτό και η τρομοκρατία ε, αποτελεί ένα μεγάλο κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς προκαλεί ε, σημαντική πηγή εξόδων και δαπανών. Ε, ακριβώς γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να αποτελέσει έναν χώρο ε, ευημερίας και ειρήνης. Γι' αυτό και ε, πρέπει να υπάρξει μια αναλογικότητα όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ο κύριος Βαγκόλη Γκόη μας μίλησε ήδη για το κόστος της απουσίας της Ευρώπης όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιέγραψε κάποιες από τις δυνητικές δράσεις που μπορούν να ληφθούν σε Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεραστούν τα κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να ποσοτικοποιήσω λίγο τους, ε, τις, τις επιπτώσεις της τρομοκρατίας και των αντιτρομοκρατικών μέτρων που λαμβάνονται. Κάναμε λοιπόν μια μεγάλη αναθεώρηση σχετικών ε, εγγράφων και οικονομικής βιβλιογραφίας. Λάβαμε υπόψη μας και δευτερογενή στοιχεία όπως είναι η, βάση δεδομένων, η παγκόσμια βάση δεδομένων για την τρομοκρατία, όπου καταγράφονται όλες οι τρομοκρατικές επιθέσεις από το 2070. Ε, έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε μια μοντελοποίηση για να καταλάβουμε καλύτερα τον αντίκτυπο της, τον αντίκτυπο της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα στην ανάλυση μας εξετάσαμε έξι τομείς ε, αντικτύπου. Πρώτον στον άνθρωπο, όσον αφορά την απώλεια ζωής και τραυματισ... τους τραυματισμούς. Δεύτερον, η τρομοκρατία έχει και φυσικό κόστος σε περιουσιακά στοιχεία και σε υποδομές. Μπορεί επίσης να έχει οικονομικές επιπτώσεις απώλειες ΑΕΠ και οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι ότι η τρομοκρατία έχει και ψυχολογικές επιπτώσεις όσον αφορά την ικανοποίηση από, το, από τη ζωή, την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εξετάσαμε και τις δημόσιες δαπάνες που ε, μπορούν και αυτές με τη σειρά τους να επλήξουν αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη. Και Επίσης εξετάσαμε τις ε, επιπτώσεις των αντιτρομοκρατικών μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι η ιδιωτικότητα, ε, και τις ελευθερίες των ατόμων. Και προσπαθήσαμε να ποσοτικοποιήσουμε, να μετρήσουμε συγκεκριμένα τις επιπτώσεις αυτές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν το, το, το, το, το, τον αντίκτυπο όσον αφορά το κόστος σε χαμένες ζωές και τραυματισμούς. Από το 2004 στο 2016 ε, χάθηκαν 669 ζωές και 4.623 τραυματίες είχαμε. Και εδώ βλέπαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κόστος γι' αυτό. Λάβαμε επίσης υπόψη μας το κόστος ε, άμεσα που πλήττει τους, ε, τα, τα θύματα, ιατρικές δαπάνες, ε, αποκατάστασης αλλά και ψυχολογικού τραύματος που προκαλείται. Ε, πέραν από αυτές τις ανθρώπινες επιπτώσεις, η τρομοκρατία έχει ε, επιπτώσεις αρνητικές στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποδομές. Συνολικά λοιπόν υπολογίσαμε ότι οι ζωές ε, οι απώλειες ζωών μάλλον ανέρχονται σε κόστος 4,3 δισεκατομμύρια ζωή την περίοδο 2004-2016 ε, το κόστος των ε, τερματισμών 0,3 δισεκατομμύρια και στην, στα περισσότερα στοιχεία 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα περισσότερα από αυτά τα κόστη προέρχονται από την περίοδο 2013-2016. Εκεί οι νεκροί ήταν ανέρχονταν σε κόστος δηλαδή ε, στα 2,4 δισεκατομμύρια, 0,1 δισεκατομμύρια και 0,1 δισεκατομμύρια πάλι όσον αφορά τις ζωές, τους τραυματισμούς και τα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν διάφορες διαδρομές για το πώς η τρομοκρατία μπορεί να ε, ε, επηρεάσει την οικονομία και την κοινωνία. Όπως σας εξήγησα, η τρομοκρατία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο ε, στην παραγωγικότητα, στην παραγωγή, και στο κεφάλαιο, στην εργασία. Μπορεί να επηρεάσει την κατανοητική συμπεριφορά ε, των ατόμων και μπορεί να επλήξει τον ε, τουρισμό, τις μεταφορές και το λιανεμπόριο. Επίσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις μειώνοντας τα κίνητρα για άμεσες επενδύσεις, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις επενδύσεις αυτές. Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι η τρομοκρατία μπορεί να διαταράξει και το διεθνές εμπόριο. Όπως για παράδειγμα γίνεται με την εισαγωγή συνοριακών ελέγχων ε, και την αύξηση μη δασμολογικών εμποδίων. Επίσης, η τρομοκρατία αυξάνει τις κρατικές δαπάνες ε, στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, κάτι που βεβαίω οδηγεί σε αύξηση των φόρων, του ελλείμματος και που προφανώς πρόκειται για χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αν, απουσία της τρομοκρατίας για άλλους τομείς όπως είναι η έρευνα και η ανάπτυξη. Από τη μακροοικονομική μας ανάλυση λοιπόν ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ε, η τρομοκρατία από το 2004 έως σήμερα είχε ε, ως αποτέλεσμα απώλεια 180 δισεκατομμυρίων ευρώ ε, απώλεια στο, για το ΑΕΠ. 358 ευρώ κατά δηλαδή. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το ποσό, το ποσό αυτό αν το εξετάσει κανείς την περίοδο 2013-2016. 87 δισεκατομμύρια όσον αφορά το, το ΑΕΠ ή 175 ευρώ κατάτομο. Επίσης, η τρομοκρατία μπορεί να έχει και πολύ σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις ε, στην ψυχολογία του πληθυσμού. Όπως ανέφερα, μέσω της μαζικής ε, κάλυψης από τα μίσα μαζικής ενημέρωσης, πολλοί άνθρωποι πλήττονται και επηρεάζονται από τις τρομοκρατικές επιθέσεις πέραν των άμεσων ε, των θυμάτων και πολλές φορές οδηγούνται οι άνθρωποι σε αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οι έρευνε μας ε, επίσης δείχνουν ότι η τρομοκρατία επηρεάζει αρνητικά την ευτυχία, την ικανοποίηση από τη ζωή και την εμπιστοσύνη ε, που δείχνουν οι άνθρωποι στους ε, θεσμούς του πολιτικούς. Και έτσι και η ψυχολογία του πληθυσμού είναι ένα τομέα ο οποίο δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς. Πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω γιατί ήταν πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο βεβαίως να αποδώσει κανείς σε συγκεκριμένες αξίες αυτές τις επιπτώσεις. Πέραν από τις ε, άμεσες επιπτώσεις ε, της τρομοκρατίας λοιπόν, μεγάλο ποσό ε, οδηγείται και κατευθύνεται και στα αντιτρομοκρατικά μέτρα που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα το 2017 ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός προέβλεψε περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ για θέματα ασφάλειας και ηθαγένειας και το, οι νέες προτάσεις για το ΠΔΠ 2021-2027 προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις. Το, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα υπερδιπλασιαστεί από το 1 δισεκατομμύριο στα 2,5 δισεκατομμύρια. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο ενωσιακός προϋπολογισμός αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα των συνολικών δεπανών που πραγματοποιούνται σε επίπεδο κράτο μέλους. Παρ' αυτά είναι πολύ δύσκολο να απολογιστούν οι δαπάνες ή αντιτρομοκρατικέ σε επίπεδο ε, κράτους μέλους γιατί τα στοιχεία αυτά συνήθω δεν, δημοσιεύονται. Παρ' αυτά εκτιμούμε ότι τα κράτη-μέλη ε, ακολουθούν παρόμοια τάση με τις ε, Ευρωπαϊκής, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτιμούμε λοιπόν ότι συνολικά οι, συνολικοί, οι συνολικές δαπάνες ε, για αντιρρομοκρατικά μέτρα ε, υπερβαίνουν τα 8 δισεκατομμύρια ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο κρατών μελών βεβαίως. Βεβαίως μια προσοχή αντιμετωπίστε αυτούς τους ε, αριθμούς που σας δίνω γιατί όπως είπα κάναμε πολλές υποθέσεις για να καταλήξουμε. Λοιπόν, τα αντιτρομοκρατικά μέτρα πράγματι είναι ένα από του βασικότερου τρόπου αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, αλλά και τα ίδια αυτά μέτρα μπορούν να ε, έχουν αρνητικέ επιπτώσει στην κοινωνία και στην οικονομία, όπω είπα για του ελέγχου στο αεροδρόμιο, που είναι ένα πολύ απτό και εύληπτο παράδειγμα. Επίση, Υπάρχουν και άλλα μέτρα που λαμβάνονται, όπως είναι οι εκδόσει, η παράνομη κράτηση, τα βασανιστήρια, η μαζική παρακολούθηση, η, η ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά μπορεί να έχουν ε, καταστροφικές συνέπειες στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, η υπερβολική ή παράνομη κράτηση ε, δε ε, πιθανών υπόπτων για εγκλήματα τρομοκρατίας μπορούν, μπορούν επίσης να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την υγεία των ατόμων αυτών, την, τις ευκαιρίες τους στην απασχόληση κτλ. κτλ. Επιπλέον, προγράμματα για την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης πολλές φορές μεροληπτούν εναντίον συγκεκριμένων θρησκευτικών ή εθνοτικών κοινοτήτων. Και αυτό πολύ συχνά επηρεάζει αρνητικά και τις ε, προοπτικές απασχόλησης των ατόμων που συμμετέχουν ή εντάσσονται σε τέτοιου προγράμματα. Όλα αυτά σας τα έχουμε άλλωστε παρουσιάσει και σε προηγούμενες μελέτες μας ε, στην Επιτροπή σα. Η έρευνά μας λοιπόν δείχνει ότι η τρομοκρατία έχει σημαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στα άτομα μέσω της απώλειας ζωής και των ε, τραυματισμών. Ωστόσο, οι επιθέσεις που έγιναν την τελευταία δεκαετία είχαν σημαντικότατες οικονομικές επίσης επιπτώσεις ε, στο ΑΕΠ συγκεκριμένα. Και εδώ ε, πρέπει να σημειώσω ότι ο αριθμό που σα έδωσα ενδεχομένω να είναι και πολύ ψηλότερο, γιατί δεν έχουμε ακόμα ε, αποδώσει σε συγκεκριμένε νομισματικέ αξίε το, το κόστο των ψυχολογικών επιπτώσεων που έχει η τρομοκρατία στους πληθυσμούς της Ευρώπης. Επίσης, τα αντιτρομοκρατικά μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις ε, είναι σημαντικά, έχουν κόστος, θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα γιατί πολλές φορές μπορούν από κοινωνική και, ε, και ε, οικονομικής άποψης να πλήξουν σοβαρά τα άτομα εναντίον των οποίων στρέφονται γεγονό πάντω είναι ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα για να καταλάβουμε ε, ε, καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος ε, τις επιπτώσεις που έχουν οι δαπάνες που λαμβάνονται σε σχέση με τα αντιδρομοκρατικά μέτρα. ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να χτίσουμε πάνω σε αυτό γιατί η πρώτη μου αντίδραση είναι κάτι για το γενικό. Οι πραγματικές επιπτώσεις εξετάζονται σε, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενική κοινωνική και οικονομική επίπτωση. Εμάς Όμω εδώ στη Λίμπη μα ενδιαφέρει να ξέρουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία του δικού μας έργου. Θα θέλαμε περισσότερες λεπτομέρειες δηλαδή. Έχω περισσότερες ερωτήσεις για το δεύτερο, τη δεύτερη παρουσίαση. Η πρώτη είναι ενδιαφέρουσα, αλλά είναι πράγματα που και εθνικοί βουλευτές μπορούν να τα ρωτήσουν για τις επιπτώσεις του, της τρομοκρατίας στην κοινωνία. Καλά, αργότερα θα υποβάλω τις ερωτήσεις μου, θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Πάντως είναι ε, ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις αυτές. Η Ναταλή που προεδρεύει, η Ναταλή Κρίσμπερ που προεδρεύει τη ειδική μας Επιτροπής για την Τρομοκρατία. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ Κλοντ. Κάποιες παρατηρήσεις πρώτα και μετά δύο ερωτησούλες. και μετά μάλιστα από αυτά που είπε και ο Προεδρός μας, ε, σας ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίασή σας, την πλήρη, τεκμηριωμένη και που προσπαθεί να δώσει κάποια στοιχεία ε, όσον αφορά την ευρωπαϊκή κοινωνία, ξέροντας ότι σε κάποιες χώρες έχουμε δεδομένα, σε κάποιες χώρες δεν έχουμε, ε, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε, όλες τις αναλύσεις πάντα. Οπότε είναι περίπλοκη η δουλειά αυτή που κάνατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Κυρίως για την ιδέα αυτή της προστιθέμενης αξίας της Ευρώπης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τόσο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όσο και στην Ειδική Επιτροπή Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεργαζόμαστε με τις εθνικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια και επιμένουμε ξανά και ξανά ότι πρέπει να αναλύσουμε και να βρούμε λύσεις σε αυτή την πρόκληση που επηρεάζει όλες μας τις κοινωνίες, όλες τις χώρες μας, τόσο τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να σας πω ότι δεν είχα το χρόνο να διαβάσω λεπτομερώς αυτά που μας στείλατε, ήμουνα και διακοπές. Οπότε δεν τα έχω αναλύσει όλα σε βάθος, αλλά εσείς υπογραμμίσατε το κόστο που είναι πάνω από 400 στο ΑΕΠ, που είναι τεράστιο ποσό. Και τα νούμερα αυτά δεν μπορούν βέβαια να αντικατοπτρίσουν με ακρίβεια το κόστος, ε, τις συνέπειες, τις ψυχολογικές, πάνω στην κοινωνία, πάνω στα άτομα, πάνω και στην ε, πολιτική γνώμη στις διάφορες χώρες. Θα μπορούσα για ώρες να μιλάω για αυτά. Πάντως έχω και δύο ερωτήσεις για τον προπολογισμό μετά από την ανάλυση που μας κάνατε όσον αφορά τις δαπάνες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εσείς πιστεύετε ότι φτάνουν τα ποσά αυτά, πιστεύετε ότι είναι λίγα. Κάνουμε πολλοί προσπάθειες να αποδώσουν τα χρήματα αυτά περισσότερο αναπτύσσοντας ε, συστήματα συλλογής δεδομένων που είναι αναγκαία για την ανταλλαγή πληροφοριών και για να μπορέσουμε τελικά να δώσουμε απαντήσεις για την πρόληψη. Έχετε αξιολογήσει λοιπόν και εκτιμήσει αυτές τις ανάγκες. Και δεύτερον, μιλήσατε για πολύ για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Μιλήσατε για την δημιουργία ενός συστήματος ε, παρακολούθησης, αντίστοιχο με αυτό των πολιτείων Εσείς τι θα λέγατε για ένα τέτοιο πρόγραμμα, ε, καθαρά ευρωπαϊκό όμως. Ευχαριστούμε, Ναταλή. Η... Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά τώρα, γιατί εξακολουθώ να είμαι διακοπές και μάλλον συγκεντρώνομαι καλύτερα στην μητρική μου γλώσσα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις εκθέσεις που μας παρουσίασαν και τους ευχαριστώ που εξέτασαν όχι μόνο την οικονομική πτυχή των επιπτώσεων της τρομοκρατίας αλλά και τις άλλες πτυχές των τρομοκρατικών επιθέσεων αλλά και το κόστος που, ε, επιφέρουν η λήψη, που επιφέρει η λήψη αντιτρομοκρατικών μέτρων. Τους ευχαριστώ επίσης για την επισήμανση ότι κάθε μέτρο στην πλειάδα τους αυτοί ε, συνοδεύονται πάντοτε από τον κίνδυνο να περιοριστούν οι θεμελιώδεις ελευθερίες, ελευθερίες και μάλιστα τη στιγμή που ακριβώς από αυτό που θέλουμε να προστατεύσουμε από την τρομοκρατία είναι οι ελεύθερες και ανοιχτές κοινωνίες μας. Θυμάμαι δε ότι Λίγο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες ε, βρέθηκα εδώ στο αεροδρόμιο και σε σιδηροδρομικό σταθμό και μιλώντας με πολίτες ε, που ζουν εδώ στην, ε, στις Βρυξέλλες μου έλεγαν ότι εμείς συνειδητά θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στα μέρη αυτά, στο αεροδρόμιο και θα παίρνουμε το μέτρο, γιατί δεν δεχόμαστε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Γι' αυτό και σε πολιτικό επίπεδο πολλέ φορέ ασκείται η πίεση να λαμβάνονται γρήγορα μέτρα, χωρίς ωστόσο αυτά να υλοποιούνται ε, όσο γρήγορα χρειάζεται ε, ή αναμένεται. Λαμβάνονται λοιπόν πολλέ φορέ μέτρα τα οποία δεν αξιολογούνται επαρκώ ούτε εκ των προτέρων αλλά ούτε και εκ των υστέρων. Γι' αυτό και χρειάζεται συνεργασία, όχι μόνο στα τεχνικά μέτρα, χρειάζεται συνεργασία στην αξιοποίηση, στην αξιολόγηση, στη συνεργασία στον ε, τομέα της καταπολέμησης τρομοκρατίας και πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι η απροθυμία να συνεργαστούν συγκεκριμένες αρχές αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλές φορές και διαφορετικές παραδόσεις τόσο στις αστυνομικέ αρχές όσο και στις δικαστικές αρχές και είναι δύσκολο να χτιστεί εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών αρχών μεταξύ των κρατών μελών και γι' αυτό και εδώ χρειάζεται πολλή δουλειά να γίνει ακόμη. Επίσης θέλω ακόμη να πω ε, κάτι για την πρόληψη και την απορριζοσπαστικοποίηση. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι η πανάκερη, η μοναδική έννοια που θέλουμε, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, προσπαθούμε μάλλον να βρούμε μία πανάκια για να, να καταπολεμηθεί η ριζοσπαστικοποίηση. Δεν υπάρχει όμως πανάκια, δεν υπάρχει μία λύση, γιατί οι καταστάσεις που επικρατούν στις διάφορες πόλεις και στις διάφορες χώρες είναι διαφορετικές. Όσον αφορά την απορριζοσπαστικοποίηση, ε, νομίζω ότι πολλές φορές δεν λαμβάνουμε επαρκή μέτρα πολύ συχνά συγκεντρωνόμαστε, επικεντρωνόμαστε σε κάποιους που είναι δυνάμει ριζοσπαστικοποιημένοι, που ενδεχομένως έχουν σχέση και με το μικρό έγκλημα, αλλά θέλω να επισημάνω και έναν άλλο, μια άλλη πληθυσμιακή ομάδα, εκείνων που επιστρέφουν ε, και όχι μόνο εκείνων που επιστρέφουν, αλλά και των οικογενειών τους και των παιδιών τους, που είναι και θύματα βέβαια, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν ενδυνάμει και δεν αρκεί να τους παρακολουθούμε αυτούς ως προληπτικό μέτρο, βεβαίως. Το ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ είναι τι εφόδια δίνουμε σε αυτά τα παιδιά ή θα δώσουμε σε αυτά τα παιδιά προκειμένου να ε, αναπτύξουν μια διαφορετική κοσμοθεωρία, μια διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο και εδώ νομίζω ότι ακόμη δεν έχουν γίνει ε, πολλά πράγματα, ούτε αρκετά. Και Τέλος, ένα ζήτημα που με απασχολεί είναι ε, το εξής. Ποια, ποια είδη ριζοσπαστικοποίησης ε, δημιουργούνται και εμφανίζονται πέραν της ε, τρομοκρατίας. Διότι εγώ τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία διαπιστώνω μια ολοένα και μεγαλύτερη προθυμία για τη διάπραξη βίαιων πράξεων και εγκλημάτων διαπιστώνουμε πέραν από τη τρομοκρατίας, ε, πέραν της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας δηλαδή, ότι υπάρχουν και άλλα εξτρεμιστικά ρεύματα, ακροαριστερά και ακροδεξιά. Υπάρχουν ε, επιθέσεις ε, σε κέντρα ασύλου, σε κέντρα παροχής βοήθειας σε πρόσφυγες, ειδικά στην Ανατολική Γερμανία μάλιστα Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, υπήρξε και ένας όχλος ο οποίος ε, ε, επιτέθηκε σε πρόσφυγες και δεν ε, σταμάτησε ούτε μπροστά στις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι λοιπόν μια, ένα δυναμικό το οποίο δημιουργείται και το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Αντί όμως να καθόμαστε να τα συζητάμε εδώ, έστω και με τον πιο συναισθηματικό τρόπο, νομίζω ότι το ζητούμενο εδώ για μας είναι να δούμε αν ε, ε, ε, λαμβάνονται επαρκή μέτρα ή αν σχεδιάζονται για το μέλλον επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών της βίας και της ριζοσπαστικοποίησης, εν γέννη πέραν της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Και αν θεωρείτε κι εσείς ένα ερώτημα προς εσάς, αν θεωρείτε ότι πρέπει αυτές οι πτυχές να ληφθούν υπόψη στη χάραξη πολιτικής από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Η Μάιτε como española. Ευχαριστώ. Μια που είμαι Ισπανίδα, με ενδιαφέρον πάρα πολύ αυτά που είπατε. Για τη μελέτη αυτή αξιολογεί αναχώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το κόστος, το ανθρώπινο, το οικονομικό, βάσει του ΕΠ, της τρομοκρατίας, πώς επηρεάζει αυτή δηλαδή την οικονομία, αλλά και την ψυχολογία των ανθρώπων στις χώρες μας και η χώρα μου έχει πληρώσει μεγάλο κόστος για την τρομοκρατία η Ισπανία. Βέβαια στη μελέτη σας φαίνεται ότι για τη Γαλλία το κόστος μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ήταν πολύ μεγάλο από πλευρά ανθρώπινων ζώων αλλά και οικονομίας. Και είναι πολύ ενδιαφέρον για το έργο της Επιτροπής μας, αυτά που λέτε, και για τις συστάσεις στις οποίες θα καταλήξει η Ειδική Επιτροπή για την Τροποκρατία. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, γιατί θα μπορέσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δίνεται στις δικές μας συστάσεις. Τώρα, τα κενά που μας βοηθάτε να καλύψουμε επίσης είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για την ειδική μας επιτροπή. Πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο έργο μας, πιο αποδοτικοί το κόστος, το συγκριτικό, πόσο στοιχίζει η τρομοκρατία και πόσο στοιχίζει το κόστος αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη δουλειά μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που θα ήθελα να προτείνω, να προσθέσω για μελλοντικές μελέτες. Το ένα είναι ότι αν με σχετικούς όρους συγκρίνουμε το 2004 και το 2013 τι έγινε στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες χώρες, με το Αφγανιστάν, με το Πακιστάν, ή με τις λεγόμενες αποτυχημένες χώρες εξαιτίας του βίαιου φανατισμού που και μας μας πλήττει, αλλά πολύ λιγότερο από ότι το Ιράκ και τη Συρία. Θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη πολύ ενδιαφέρουσα που να συγκρίνει το κόστος αυτών των φανατικών ιδεολογιών και πόσο κοστίζει το να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία ένα, μια χώρα η οποία είναι λεγόμενα αποτυχημένη χώρη, fail state, ε, φυσικά και έχει τεράστιο κόστος εξαιτία αυτού. Στην Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, μια από τις τελευταίες παρεμβάσεις που ακούσαμε ήταν από έναν ε, ειδικό για την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, μας μίλησε για το Ισραήλ και για την σημαντική τεχνολογική επένδυση που κάνουν οι Ισραηλινοί και πώς αυτό αποδίδει. Γιατί είναι πολύ αποτελεσματικό στην καταπολέμηση ακριβώς ε, διάφορων εγκληματικών απειλών αλλά και πόσο αποδίδει οικονομικά το γεγονό ότι μπορούν να πουλήσουν αλλού τη δικιά του τεχνολογία, αυτή που έχουν αυτή αναπτύξει για την καταπολέμηση τη τρομοκρατίας. Μπορείτε να μα μιλήσετε λίγο για αυτέ τι δυνατότητε. που βοηθούν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε συνάδελφοι. Μην ξεχνάμε και το χρόνο, να είμαστε σύντομοι. Ο κύριος Κάρσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με διάφορα φαινόμενα. Σε επίπεδο, όλοι έχουμε έχουμε μια νέα χάρτα που λέει ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να νιώθουν ασφαλείς. Αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να σταθμίζεται καλά. Να δούμε δηλαδή ότι ο περιορισμός των δικαιωμάτων για να τους προστατεύουμε πρέπει να είναι περιορισμένος και αυτός. Να είναι λίγος ο περιορισμός των δικαιωμάτων τους. Τώρα σε μια κατάσταση τρομοκρατικής απειλής η κοινωνία συμφωνεί για τον περιορισμό των δικαιωμάτων της. Αυτό γίνεται. Αργότερα όμως δεν ε, ξέρουμε πώς να αποσύρουμε τους περιορισμούς αυτούς. Οι αρχές διστάζουν, δεν θέλουν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση γιατί φοβούνται. για περισσότερο ψυχολογικούς λόγους, γιατί τελικά αυτά τα μέτρα δεν καταπολεμούν την τρομοκρατία, απλώς πείθουν την κοινωνία ότι οι αρχές έτσι καταπολεμούν την τρομοκρατία. Παράδειγμα, αυτό που έγινε στη Γαλλία με την έκτακτη νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας, όπου αποσύρθηκε αργότερα, αλλά φάνηκε ότι το 90% πέρασε στην κανονική νομοθεσία και όχι στην έκτακτη. Τα μέτρα λοιπόν που λαμβάνονται πρέπει να είναι αναλογικά και να βλέπουμε κάθε τόσο είναι αναγκαίες αυτές οι λύσεις. Άλλο παράδειγμα, ασφάλεια στα αεροδρόμια. Στην αρχή, μετά την επίθεση του 2011, την τρομοκρατική, απαγορεύτηκαν τα υγρά, η μεταφορά υγρών στο αεροπλάνο δεν είναι αναγκαίο. Δεν έχει νόημα. Εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλού δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Δεν επηρεάζει καθόλου την ασφάλεια των επιβατών ένα τέτοιο μέτρο. Αλλά κάποιοι κερδίζουν χρήματα από αυτό. Τα αεροδρόμια. Διότι ο κόσμος αγοράζει τελικά νερό, δεν το παίρνει από το σπίτι του, το αγοράζει στο αεροδρόμιο αφού έχει περάσει τον έλεγχο. Άρα κερδίζουν από αυτό. Οπότε, για να συνοψίσω, πιστεύω ότι όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, Πρέπει να προστατεύουμε και το δικαίωμα στην ασφάλεια βέβαια των ανθρώπων που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας κάθε φορά που κάνουμε τεχνολογικές προσαρμογές, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε τόσο τα μέτρα αυτά πρέπει να τα αναθεωρούμε, να τα ξανακοιτάμε, να τα αξιολογούμε, είναι όντω αναγκαία ή περιορίζουν τελικά υπερβολικά την ελευθερία και τα δικαιώματα των πολιτών. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Κέγγι είναι μετά η κυρία Σαρτζεντίνη, ο κύριος Ντεπρέ και η κυρία Στίβενς. Και εδώ κλείνει ο κατάλογος ομιλητών. Εντάξει, δύο λεπτά το πολύ παρακαλώ καθένας. Συμφωνεί. Σεσίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τους ε, εμπειρογνώμονές μας για τις παρουσιάσεις τους. Και ήθελα να κάνω και εγώ κάποια σχόλια και μερικέ ερωτήσει. Από τη μελέτη προκύπτει ότι η τρομοκρατία είναι μια από τι βασικέ ανησυχίε των Ευρωπαίων πολιτών. Και αυτοί θέλουν μέτρα. Θέλουν οι κυβερνήσει να αναλάβουν περαιτέρω μέτρα. Όμω οι δαπάνε για τα μέτρα κατά τη τρομοκρατία αυξάνονται σε όλα τα κράτη-μέλη. Και βεβαίω είναι προφανεί οι δυσκολίε. Από την αρχή τη παρουσίαση φάνηκε ότι οι κυβερνήσει δεν έχουν ε, ε, Ευκολία στο συντονισμό των ε, διοκτικών τους αρχών. Ε, δεν υπάρχει σεβασμός θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συντονισμός μεταξύ των υπευθύνων αρχών. Είναι μη ικανοποιητικό αυτό που συμβαίνει. Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνε τους ενώπιον των πολιτών. Το σημείο που θέλω να τονίσω και αποτελεί μέρος και της παρουσίαση που κάνατε όταν μιλήσατε και για τις ψυχολογικές επιπτώσεις ε, στους, στον πληθυσμό, στους πολίτες. Αναρωτιέμαι Εάν σκεφτήκατε οι ανακοινώσει, οι πληροφορίε και το πώ παρουσιάζονται, τι επιπτώσει μπορεί να έχουν. Το τι λέει ο τύπο δηλαδή και οι ειδήσει. Πολλέ φορέ υπάρχουν ψευδείς ειδήσει. Και αυτό ε, πολλέ φορέ τροφοδοτεί την τρομοκρατία. Αυτό έχει και μια ψυχολογική ε, πτυχή, διότι εκτό που επηρεάζει συγκινησιακά του πολίτε, έχει και οικονομικέ επιπτώσει. Όποιο ε, προβάλλει ψευδείς ειδήσει, σκοπό έχει κάτι να κερδίσει. Και να τελειώσω σε κάτι άλλο, λέγοντας κάτι άλλο, πάλι για την επικοινωνία και την ε, προβολή των νέων. Μπορεί κανείς να χειραγωγήσει, να ε, χρησιμοποιήσει τα νέα και τις ειδήσει για να επηρεάσει και τη χάραξη της πολιτικής. Το τελευταίο που ήθελα να σχολιάσω είναι αν ε, αποτιμήσατε το κόστος για τις οικογένειες των θυμάτων ή κάποιες ομάδες του πληθυσμού, με τι προληπτικά μέτρα μπορούσαμε να αποφύγουμε να, τα κάνουν, να τους κάνουμε να αισθάνονται θύματα. Οι οικογένειες αυτές που σε μια κοινωνία δεν έχουν δουλειά, ε, μπορεί να βρεθούν στη θέση του θύματος σε μια δεύτερη φάση, λόγω επιλογών που δεν έχουν κάνει οι ίδιοι απευθείας. Ευχαριστώ. Κύριε Σαρχεντίνη. Κύριε Φανπαλεχόη, ξεκινήσατε την παρουσίασή σας λέγοντας ότι αν ψάχνουμε και επιχειρηματολογία στα κράτη-μέλη να πούμε ότι είναι ζωτική σημασία ε, η αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας, ε, υπάρχει πάντα το αντεπιχείρημα ότι κοστίζουν πολύ τα μέτρα. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι χώρες μέλη θέλησαν να επιβάλλουν νομοθεσία για την οποία εξακολουθούμε να έχουμε αμφιβολίες, το PNR για παράδειγμα, και κοστίζει. Ακολουθώ την επιχειρηματολογία σας, αλλά θέλω να καταλάβω τι είδους πολιτικές θα προτείνατε εσείς να ακολουθήσουμε με την επιχειρηματολογία αυτή για το πόσο κοστίζει η απουσία της Ευρώπης, γιατί όσα κοστίζουν για την προστασία των ε, δεδομένων, κοστίζουν πολλά, αλλά έχουν περάσει με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία από τις χώρες μέλη. Ευχαριστούμε κύριο Δεπρέ. Ζεράρ. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Ναι. Μια ερώτηση μετά από τα όσα ακούσαμε. Ο τίτλος της έκθεσης, υποτίτλος τέλο πάντων, είναι κόστος της αποσίας της Ευρώπης. Cost of non-Europe. Άκουσα την ε, αξιολόγησή σας, πόσο στοιχίζει δηλαδή στις χώρες μέλη, πόσο στοιχίζει στους ιδιώτες, αλλά εγώ δεν βρήκα αυτό το κόστος της απουσίας της Ευρώπης. Είδα ποιο είναι το κόστος της τρομοκρατίας Δηλαδή, αν πρέπει να δικαιολογήσω στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη τα χρήματα τα οποία θα βάλουμε σε κάποιο σύστημα που θα δημιουργήσουμε, θα ήθελα να ξέρω αν η κάθε χώρα από μόνη της αναλάμβανε την αντιμετώπιση αυτή, ποια θα ήταν η διαφορά, πόσο θα κόστιζε παραπάνω. Τελικά, δεν κάνατε μια παρουσίαση για το κόστος της απουσία τη Ευρώπης, αλλά για το κόστος της Τρομοκρατία μέσα στην Ευρώπη. Κάνω λάθο. Ε, και υπάρχει, ήταν και μια από τις ερωτήσεις μου. Η κυρία Στίβενς, η τελευταία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι συνεισηγήτρια της έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ λοιπόν τους ερευνητές για τις παρουσιάσεις τους και για τη συζήτηση όσον αφορά την τρομοκρατία και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Πρόκειται για ένα ευρύ πεδίο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ. την έκθεση αυτή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε ώστε να προχωρήσουμε στην εκπόνηση της έκθεσής μας με τροπολογίες και στο τέλος χρονιάς ελπίζουμε ότι θα την έχουμε. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στην ασφάλεια και τα δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντική, πρέπει να την προστατέψουμε. Είναι δύσκολο βέβαια να βρεθεί αυτή η σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Και αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και θα έχουμε και στο μέλλον. Οι κυβερνήσεις, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, οι αρχές, όλοι. Ούτε πρέπει να στιγματίζονται κάποιες ομάδες. Σίγουρα κάποιες ομάδες μπορεί να είναι πιο επικίνδυνες από άλλες, αλλά υπάρχουν πολλές μορφές τρομοκρατίας. Και δεξιά και αριστερά. Και όλες αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη σωστή ισορροπία. Επίσης, υπάρχει μεγάλη πρόκληση μεταξύ των χωρών μελών κάποιες αστυνομικές υπηρεσίες, Η δικαστικές, έχουν μια διαφορετική νοτροπία, παραδόσεις και πρέπει να υπάρξει καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους πολίτες. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη είναι τελικά αυτοί που πρέπει να κοιώνται την ασφάλεια. Και αυτοί είναι που πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει καλή συνεργασία. Επίσης, καλή συνεργασία πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις εθνικές αρχές και τις ευρωπαϊκές, Europol, Eurojust. Όλοι έχουν να προσφέρουν κάτι. Οι κυβερνήσεις όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουν ό,τι ήδη υπάρχει να κάνουν χρήση αυτών. Και βέβαια υπάρχει και σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα. Δεν θα πρέπει η Ευρώπη να αντικαθιστά τις εθνικές αρχές. Σε πολλές περιπτώσεις όμως έχει αποδειχτεί η αξία της καλής συνεργασίας, που όμως δεν υπάρχει πάντα. Και πρέπει και αυτό να υπολογιστεί στο κόστος της απουσίας της Ευρώπης. Όντω λείπει το κόστος της απουσίας Ευρώπης. Εγώ αυτό θα ήθελα να ξέρω. Ποιο είναι το κόστος της απουσία της Ευρώπης. Συμφωνώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί το ότι έχει γίνει μέχρι τώρα, δηλαδή ποια μέτρα έχουν λειτουργήσει καλά, ποια αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και ποια όχι. Αυτό θα βοηθήσει και μας στην έκθεσή μας. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Είναι λογικό οι παρουσιάσεις σας να δημιουργούν τέτοιες συζητήσεις και απορίες. Πολύ σύντομα έχω μια ερώτηση κι εγώ και εσείς θα απαντήσετε. Είναι λίγο πολύ αυτό που είπε και ο κύριος Ντεπρέ για μας, για την Επιτροπή μας Λίμπε. Που γνωρίζουμε ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιούμε τώρα το ΣΥΣ2, το εισαγγελικό ένταλμα, η Europol, που φαίνεται ότι πάει καλά. Η ερώτηση μου είναι, ποια είναι η αντίληψη για την προστιθέμενη αξία. Εσείς στην έρευνά σας μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η αντίληψη για αυτήν την προστιθέμενη αξία στο Συμβούλιο, για παράδειγμα, μιλάμε για το PNR, δεν το εφαρμόζουν. Είναι μια εντελώ διαφορετική αντίληψη αυτή που έχουν οι χώρες μέλη σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εμείς σαν προστιθέμενη αξία. Εσείς μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό κόστος. Πριν περάσουμε σε άλλα μέτρα για τον κυβερνοχώρο, λειτουργότητα κτλ. θα πρέπει αυτό να ξέρουμε. Για να απαντήσετε. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Να συγχαρώ τον, να ευχαριστήσω μάλλον τον ε, κύριο Ντεπρέ, διότι η μελέτη αυτή για το κόστος της απουσίας της Ευρώπης δεν έχει ολοκληρωθεί και απολύτως. Και αυτό διότι ξεκινάμε με το θέμα πρόληψη, προστασία, εμ, εντοπισμός και εμ, δίωξη. Αυτά είναι τα τέσσερα πί που θέλουμε να τα δούμε σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Και η απάντησή μου είναι προφανώ όχι. Ε, χρειάζονται περισσότερα αποδεκτικά στοιχεία. Αυτό προκύπτει ω πόρισμα και από τη μελέτη. Και αυτή την απάντηση θα είχα και στο σχολείο τη κυρία Αρχεντίνη. Διότι το κόστο τη ε, έλλειψη Ευρώπη, Ευρωπαϊκή απόκριση σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι κάνουμε μεν κάτι, αλλά δεν το κάνουμε αρκετά αποτελεσματικά. Δηλαδή, να μην κάνουμε κάτι εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων κάποιων πολιτών. Αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί με τα κατάλληλα μέτρα. Και αυτό με οδηγεί και στην απάντησή μου στην κυρία Κρισπέκ, διότι μιλάμε για πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EFTU ε Πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη ποινική προσέγγιση κοινή σε αυτά τα θέματα ε, και να δούμε ποια είναι η προστεθέμενη αξία σε σχέση με το πλαίσιο που ήδη ισχύει και κατά πόσον ε, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα επιτρέπει ένα τέτοιο σύστημα να λειτουργεί. Διότι η δικονομία είναι πολύ αυστηρή προ αυτά. Και εδώ σχόλιο και για όσα είπε και η κυρία Στέιβενς. Είπατε πώ πρέπει να εξισορροπήσουμε την ελευθερία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη. Ε, χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια. Αυτό ήταν το πρώτο σα σχόλιο όμω. Ε, περισσότερη ασφάλεια θέλουμε από τα μέτρα που προτείνονται, διότι αν δεν είναι αποτελεσματικά. Τα θεμελιώδη δικαιώματα πάλι δεν επιτρέπουν να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενο σκοπό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια πραγματική, ένα πραγματικό άλμα ποιότητα εδώ. Και Μπορεί να είναι πολιτικός ε, λιγότερο ελκυστικό αυτό που θα προταθεί, όμως μας ενδιαφέρει το να έχει αποτέλεσμα στην πράξη. Από τη στιγμή της πρόληψης μέχρι τη δίωξη των ε, συγκεκριμένων προσώπων. Τώρα πάντοτε μπερδεύομαι με τους Ισπανούς ε, ευρωβουλευτές. Κυρία μου, ρωτήσατε μια, θέσατε μια πολύ εύστοχη ερώτηση και αυτό βεβαίω έχει να κάνει και με τι αρμόδιοτητε άλλων επιτροπών αυτού του σώματο, όπω των εξωτερικών υποθέσεων. Πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη στον χώρο των εξωτερικών υποθέσεων ω προ την πρόληψη τη τρομοκρατία. Στην κυρία Σίπελ θα απαντούσα το εξή. Κάτι που είδαμε στην έκθεση και ίσως και να το έχετε προσέξει και εσείς είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να κατηγοριοποιήσει καλής τον εξτρεμισμό στην τρομοκρατία σε αντιδιαστολή με τα εγκλήματα μίσους. Είναι θέμα όρων, αλλά οι πράξεις ε, δεν πάβουν να είναι βίες. Αυτό κάπως πρέπει να καλυφθεί στην όλη μας συζήτηση. Και όταν είπα ότι πρέπει να προσέξουμε να μην ε, ε παρονομάζουμε αυτό που θέλουμε να διώξουμε, ε, το στόχο των διώξεων, θα πρέπει να, είναι, να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς το στόχο των όσων σχεδιάζουμε εδώ για το κυβερνοέγκλημα. Η κυρία Κιέγγε νομίζω. Ναι, το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, το κυβερνό έγκλημα είναι θέματα που απασχολούν την Επιτροπή σας. Θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη από κοινού και να δούμε κατά πόσο η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ίσως η κορυφή του παγόβουνου ε, για πολλά πράγματα που μας απασχολούν και θα πρέπει να τα δούμε σφαιρικά. Θα σταματήσω εδώ. Και από μένα λίγες παρατηρήσεις, γιατί τα, εξήγησε πολύ καλά και ο Βούτερ, αλλά για το κόστος της απουσίας της Ευρώπης και την μελέτη αυτή από την σκοπιά ενός να Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται με την προστιθέμενη αξία εδώ. Πρέπει κανείς να δει σε κάθε μέτρο τι ε, αντίκτυπο είχε, δηλαδή τι αποφεύχθη χάρη στην έπρεξη αυτού του μέτρου. Αυτό ε, ε, επηρέασε πάρα πολύ τη μελέτη μας. Ε, δεν θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει λέγοντας ότι υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία που δείχνουν ότι η αύξηση των δαπανών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορεί να περιορίσουν το κόστος από τις μεγάλες επιθέσεις. Όμως οι τρομοκρατικές ομάδες αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν. Αν τώρα λοιπόν ξοδέψουμε πολλά για ένα συγκεκριμένο μέτρο, απέναντι αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν οργανώνουν μικρότερε κλίμακε επιθέσει. Και αυτέ δημιουργούν προβλήματα και σκοτώνουν πολλού πολίτε. Και άλλου. Δεν είναι εύκολο να το αξιολογήσει κανεί. Και βεβαίω ε, περιέχει και πολλά στοιχεία βεβαιότητα Ω προ τον ψυχολογικό αντίκτυπο. Πράγματι, τα μέσα παίζουν σημαντικό ρόλο. Ω προ τον ψυχολογικό αντίκτυπο. Βεβαίω, μέσα σε δευτερόλεπτα μπορεί κάποιο σήμερα να πέσει θύμα επίθεση και αυτό επηρεάζει μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού. Ε, πέρα από τα ίδια τα θύματα. Αλλά και εδώ τα αποδεκτικά στοιχεία διαρκώ προκύπτουν. Δεν ξέρουμε γιατί οι τρομοκρατικέ επιθέσει έχουν ε, διαφορετικό αντίκτυπο από άλλα εγκλήματα. Ξέρουμε τι ε, γνωστέ περιπτώσει ε, των Πολιτείων με τι σχετικέ βομβιστικέ επιθέσει που έδειξαν ότι η αντίδραση των ε, ανθρώπων ήταν διαφορετική σε σχέση με την ε, ε, επίθεση σε ένα δημοτικό σχολείο που πυροβολήθηκαν 20 παιδιά. Αυτό δεν επηρέασε πάρα πολύ την καθημερινότητα των πολιτών. Πρέπει να γίνουν και άλλε έρευνε λοιπόν και μελέτε εδώ για να καταλάβουμε καλύτερα τι διαφορετικέ ψυχολογικέ επιπτώσει. Σίγουρα τα μέσα μαζική ενημέρωση έχουν μια, μια σχέση που θα μπορούσαμε να την πούμε συμβιωτική με την τρομοκρατία. Πολλέ φορέ διωγγώνουν τον αντίκτυπο και την προβολή των τρομοκρατικών ομάδων. Ω προ το κόστο για τι οικογένειε και τα θύματα, και όσων βρεθούν στη θέση του θύματο. Βεβαίω, το κόστο αυτό ε, στα πλαίσια αυτή τη έκθεση δεν το καλύψαμε. Υπήρξαν όμω ε, σχετικά αποδεκτικά στοιχεία από την έκθεση για την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, καθώς και αυτήν για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι συνθήκε κράτηση, και δείχνουν ότι όσοι ε, βρίσκονται σε καταστάσεις κράτησης ακραίες, έχουν και άλλα προβλήματα μετά. Ξέρω εγώ δεν βρίσκουν απασχόληση ή μπλέκουν σε άλλα εγκλήματα και αυτό έχει ένα κόστος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε επερώτηση? Όχι. Νομίζω εδώ Εδώ το Άγιο Δισκοπότηρο της όλης αναζήτησής μας είναι η προστεθέμενη αξία των όσο κάνουμε για την ε, τρομοκρατία. Το πόσο μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις σε συγκεκριμένους χώρους και τομείς. Ποια είναι η προστεθέμενη αξία του ενός και του άλλου. Των κοινών ομάδων έρευνα, του συστήματος ΣΥΣ2, αυτό δεν απλό. Είναι τόσο δύσκολο να κάνει κανείς ε, ως πακέτο αυτή την αξιολόγηση. Προφανώς δεν είναι κριτική Γι' αυτό κάναμε και τόσο διεξοδική και εντατική συζήτηση εδώ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι για την Επιτροπή μας είναι θέμα κεντρικής σημασίας. Είναι πραγματικά για μας ε, ο κολοφόν της αναζήτησής μας. Κάποια στιγμή πρέπει να μπορούμε να τα μετρήσουμε και όλα αυτά. και στο χώρο του κυβερνού εγκλήματος που είναι μια πραγματικά έρημος από την πλευρά των στοιχείων. Δεν υπάρχει τίποτα. Ε, πρέπει να δούμε λοιπόν και τις πρακτικές επιπλοκές. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε σε αυτήν την ατραπό, διότι πραγματικά και εμείς σαν τους υπότες της τρογγυλής τραπέζης αναζητούμε το Άγιο Δισκοπότηρο. Ευχαριστώ πολύ που τα συζητήσαμε με τρόπο τόσο ευφύ όλα αυτά. Ε, σας εύχομαι καλή δουλειά ε, σε προσθήκη της ήδη καλής δουλειάς που έχετε κάνει. Και συνάδελφοι προφανώς αυτό στα προσεχώς θα το ξαναδούμε. Είναι φοβερή η δουλειά που κάνει η υπηρεσία ερευνών. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο. So colleagues, we move straight to point 10. Πάμε απευθείας στο σημείο 10, συνάδελφοι. Γνωμοδότηση για τη συνεργασία της Eurojust με την Αλβανία. Διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας, μόνο διαδικαστικά ως ΛΥΜΠΕ. Η συμφωνία ακολουθεί πιστά το πρότυπο ανάλογων συμφωνιών της Eurojust με τρίτες χώρες και τις σχετικές ρήτρε για τις θεωρήσεις ή την απελευθέρωσή τους. Θα ήθελα λοιπόν, συνάδελφοι, να σκεφτείτε κατά πόσον ε, είναι απαραίτητο να υποβληθούν εδώ τροπολογίε. Μόνο διαδικαστικέ ε, είναι δυνατόν να υποβληθούν. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το περιεχόμενο τη συμφωνία και να δώσω το λόγο στην Λάουρα, εφόσον είναι εδώ η εισηγητριά μας, η κυρία Φεράρα. Λάουρα, σε παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι καθοριστικός ο ρόλος της συνεργασίας δικαστικών αρχών μεταξύ τους για να ερευνήσουν και να προλάβουν και εγκλήματα που έχουν σχέση με την τρομοκρατία και τις οργανωμένες ομάδες εγκλήματος, οι μαφίες τα δίκτυα των εγκληματικών οργανώσεων ξεπερνούν τα σύνορα των Ευρωπαϊκών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν πολυεθνικές λειτουργούν. Πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε ε, δραστικά να καταπολεμήσουμε τη δράση τους. Βάσει των στοιχείων του ΟΗΕ και της ε, Ευρωπόλ, πολλοί είναι οι Ελβανοί μαφιόζοι που στην διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμού, ε, ξέπλυμα βρωμικού χρήματο, πορνεία, εμπορία ανθρώπων έχουν εκτενή δράση. Θα πρέπει να δούμε ότι είναι φυσική διέξοδος η Ιταλία και γεωγραφικά για την εγκληματική δράση των, αλβανικών, των αλβανών μαφιόζων προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν ε, η Ευρωπόλ και στο μέλλον να μπορέσει να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες και με άλλα τρίτα κράτη για να ενισχύσει τη δικαστική της συνεργασία. Ελπίζουμε ότι η συμφωνία αυτή θα διευκολύνει την καταπολέμηση αυτών των σοβαράτων των εγκλημάτων που είναι και επικίνδυνα και ότι θα ε, προχωρήσει αυτό προς όφελος και της Αλβανίας και των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως τώρα ε, κάποιες συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες έχουν ήδη συναυθεί μεταξύ των οποίων είπα Νορβηγία, Ελβετία, Μακεδονία. Και όλες αυτές οι συμφωνίες είναι βεβαίως ακόμα ε, καθόλου αρκετές για την πραγματική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και της θερμοκρατίας. Ελπίζω να συνεχιστούν η συνάψη συμφωνιών για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών και η αρμονική δικαστική συνεργασία. Και εν ώψη τη επιθυμία τη για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αλβανία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο προσαρμόζοντας την ε, νομοθεσία της ε, στις βέλτιστες πρακτικές και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έχει ήδη εγκρίνει νόμους κατά της μαφίας και ποινική δίωξη η Αλβανία, προκειμένου να είναι αποτελεσματική στη δράση τη και κάποια πρόοδο έχει, πρόοδος έχει επιτελεστεί και στην ε, κατάσχεση και δίμευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν αποκτηθεί από εγκληματικέ δράσει. Επίση, συνεργασία με τι αστυνομίε των κρατών μελών των τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιωθεί. Η ε, συνεργασία δικαστικών και αστυνομικών αρχών μπορεί να βελτιωθεί όμω περαιτέρω. Η συμφωνία που πρόκειται να εγκρίνει το Κοινοβούλιο θα επιτρέψει να διευκολυνθεί αυτή η συνεργασία και ελπίζουμε να έχουμε αποτελέσματα που να επιτρέψουν να εντυπωσιακοποιηθεί η συνεργασία για την καταπολέμηση του, του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος, ε, της διακίνησης των νοικοτικών και της εμπορίας ανθρώπων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φεράρα. Κύριε Τιέρ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τσεχικά. Βάλτε σας παρακολουθώ τα ακουστικά σας. Λοιπόν, ως σκιώδης του ΕΛΚ Υποστηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας να υποστηριχθεί αυτή η συμφωνία. Θα εμπλουτίσει το οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ποτέ δεν αρκούν τα μέτρα που λαμβάνονται και εδώ σημειώνουμε ότι η Αλβανία έχει σημειώσει μεγάλη προόδο και μέσω αυτής της νέας συμφωνίας Ένωσης και Αλβανίας η Αλβανία θα ενταχθεί καλύτερα και θεσμικά ε, στην ε, συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα βοηθήσει τη χώρα αυτή και την ε, προετοιμασία της χώρας αυτής για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γκρίσμπεκ. Ευχαριστώ. Σύντομα, δύο σημεία από τη δικιά μου πολιτική ομάδα. Και για μας η συμφωνία αυτή της Eurojust αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στάδιο και ως κοιόδες συζυγήτρια φυσικά και ε, καλό όλους να εγκρίνουν το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής ανάμεσα στη Eurojust και την Αλβανία. Φυσικά και χαίρομαι για αυτή τη συνεργασία με μια γείτονα χώρα για να καταπολεμήσουμε μαζί το λαθρεμπόριο, το οργανωμένο έγκλημα και κυρίως την τρομοκρατία. Αυτό μας επιτρέπει επίσης να κατανοήσουμε πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η Eurojust και αναγκαίο τη δικαστική συνεργασία που επιτρέπει την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Ελπίζω και όσον αφορά την δημοσιονομική πτυχή να εισακουστούν οι επιθυμίες της Eurojust. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε την εισηγήτριά μας. Θα πρότεινα να ακολουθήσουμε αυτά που μας είπε σε σχέση με τις προθεσμίες 31 Αυγούστου αν υπάρχουν τροπολογίες που θέλετε να καταθέσετε σχετικά με τα διαδικαστικά θέματα βεβαίως μπορείτε να το κάνετε ε, Λάουρα θέλεις να προσθέσεις κάτι όχι ωραία σε ευχαριστούμε πολύ για το έργο σου και βεβαίως και τους σκιώδεις για το δικό τους ευχαριστώ so, we now proceed. Ωραία. Οπότε περνάμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης για σήμερα που είναι το Προεδρείο καλωσορίζουμε του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Μετανάστευση. Θα έρθετε εδώ στο βήμα. Maybe maybe I can introduce the while while colleagues are coming to the front. Okay, so I'm very pleased. Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζουμε και καλωσορίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Μετανάστευσης. Για όσους δεν το γνωρίζετε, το φόρουμ αυτό ε, είναι ένα φόρουμ υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της ε, Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Κάντρι Σούβα που εκπροσωπεί το PICUM, την πλατφόρμα για τη διεθνή συνεργασία για τους ε, ε, μετανάστες χωρίς χαρτιά. Έχουμε μαζί μας επίσης την κυρία Σίλβια Τζουλίνη από την ε, οργάνωση Generation 2 for Rights, Equality and Diversity, μια μη, μη κερδοσκοπική οργάνωση που αποτελείται από άτομα με διαφορετική καταγωγή που συνεργάζονται για την ε, προώθηση της ίσης συμμετοχής σε μια ε, κοινωνία χωρίς ε, διακρίσεις. Έχουμε επίσης μαζί μας τον κύριο Άντεμ Κούμτσου από την Unity, την νέα Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων. Έχουμε μαζί μας επίσης τον κύριο Κρίστιαν Πυρβουλέσκου που εκπροσωπεί την ΕΟΚΕ που θα είναι όλοι τους στη διάθεσή μας για να απαντήσουν και στις ερωτήσεις μας. Επίσης, έχουμε μαζί μας την κυρία Λάουρα Κοράντο από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επίσης συμμετέχει και στο Προεδρείο. Τον περασμένο Ιανουάριο, λοιπόν, ε, στην Ελίμπε παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση του έργου του Προεδρείου και λάβαμε και μια παρουσίαση του έργου τους ε, βάσει των ετήσιων εκθέσεων που ε, καταρτίζονται. Η τελευταία συνεδρίαση του φόρουμ έγινε στις 6 και 7 Μαρτίου του 2018 και το θέμα ήταν προς μια πιο συμπεριληπτική αγορά εργασίας για τους μετανάστες, αξιοποίηση των δυνατοτήτων και αντιμετώπιση των προκλήσεων. Βεβαίω πρόκειται για μια πλατφόρμα διαλόγου για τη μετανάστευση και από αυτή την άποψη μας ενδιαφέρει πολύ το έργο αυτής της πλατφόρμας ως Επιτροπή καθώς μας δίνει μια άμεση εικόνα για το τι ε, θέσεις ε, υιοθετεί η κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις καθώς η πολιτική ατζέντα ε, συμπεριλαμβάνει αυτά τα θέματα σε πολύ ψηλό σημείο. Λοιπόν, Σίλβια, παρακαλώ να σου δώσω το λόγο. Έχεις πέντε λεπτά και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μέλη της Επιτροπής μας που είναι ακόμη εδώ και που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση αμέσως μετά. Σίλβια, ευχαριστώ. Καλημέρα, είμαι η Σίλβια Τζουλίνη μαζί με τον Φερνάντο Μπιάγκ εκπροσωπώ ε, τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών ε, σε αυτό το φόρουμ μετανάστευση. Ε, το φόρουμ αυτό ε, δημιουργήθηκε ε, από συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή το 2015. Ήταν ε, μια μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Φόρου Κοινωνικής Ένταξης που υπήρχε το 2009-2014. Και τα βασικά θέματα που μας απασχολούν είναι η ένταξη των μεταναστών στην αγορά και συμμετέχουν 280 εκπρόσωποι από οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και εκπροσώπους ε, των κρατών μελών, ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των τοπικών αρχών. Το φόρουμ φέτος ξεκίνησε με μαρτυρίες από δύο μετανάστες. Ο ένας επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι είναι πολύ εύκολο να φτάσει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νομίμως, αλλά και πόσο εύκολο είναι τελικά να χάσει τα χαρτιά του. Δηλαδή, καταφθάνουν άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση νόμιμα και στη συνέχεια χάνουν τα χαρτιά τους. Ο άλλος μετανάστης επικεντρώθηκε σε πρακτικές δυσκολίες, γλωσσικά εμπόδια ή δυσκολίες στο να ανοίξει κανείς τραπεζικό ε, λογαριασμό. Επίσης, με αυτές τις δύο μαρτυρίες, το φόρουμ θέλησε να τονίσει ότι είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη και οι μετανάστες στη χάραξη πολιτικής. Και αυτό ε, είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Στη συνέχεια διοργανώθηκαν εργαστήρια όσον αφορά τις δεξιότητες αλλά και την ε, εργασιακή εκμετάλλευση και την ε, πολυμορφία στον χώρο εργασίας. Στις εργασίες μας διαπιστώσαμε την ανάγκη να, συλλο... να συλλεχθούν στοιχεία σε σχέση με τις δεξιότητες. Να δημιουργηθεί από αυτά τα στοιχεία μια βάση δεδομένων, η οποία θα μας βοηθήσει στα εξή δύο πράγματα. Πρώτον, μπορεί ε, να καταγραφούν οι δεξιότητες των μεταναστών που δεν είναι πάντοτε τυπικές και ταυτόχρονα μπορεί, μπορούν και οι εργοδότες να ενημερωθούν για αυτές τις δεξιότητες, ακόμη και αν κάποιος δεν διαθέτει τυπικό παραδοσιακό βιογραφικό και παρόλα αυτά να προβεί σε πρόσληψη μετανάστη. Μια σημαντική πρόταση που ακούστηκε ήταν να αξιοποιηθούν τα ταλέντα και οι δεξιότητες σε τυπικές ε, συνθήκες. Με άλλα λόγια, μπορεί κάποιο μετανάστη να, μην να, να, να μην μπορεί να αποδείξει τα τυπικά του προσόντα, αλλά μπορεί να τα αποδείξει στην πράξη. Επίση, διαπιστώθηκε έλλειψη ενημέρωση των εργοδοτών, που δεν ενημερώνονται και δεν γνωρίζουν για τι νέε αφήξει. Ή πολύ μπορεί να μην γνωρίζει ένα εργοδότης ε, τι συμβαίνει σε σχέση με την άδεια ενό ενός ε, μετανάστη. Τονίστηκε λοιπόν η ανάγκη να υπάρχει μια προβλεψιμότητα, διότι αυτή η έλλειψη προβλεψιμότητας σε σχέση με το ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί και να εμποδίζει πολλές φορές την πρόσληψη ενό μετανάστη. Ταυτόχρονα συζητήθηκε η ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους εργοδότες να προσλαμβάνουν μετανάστες, να διοργανωθούν ε, εκπαιδευτικοί κύκλοι σε σχέση με πολιτιστική εκπαιδευτική κύκλη ε, και για τους εργοδότες αλλά και για τους μετανάστες, ώστε να γνωρίζουν ποιες ακριβώς καταστάσεις θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και περισσότεροι κανόνες. Επίσης, πρόσβαση στην δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους, ανεξάρτητα από το καθεστώς υπό το οποίο ζει κανείς και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό για να αποφεύγονται ε, περιπτώσεις εκμετάλλευσης στην εργασία. Επίσης, αυτοοργάνωση και ε, μεταξύ των ίδιων των μεταναστών ε, και ε, με διάδοση επιτυχημένων περιπτώσεων ε, και ενημέρωση και των υπόλοιπων μεταναστών για το πώς κάποιοι μετανάστες τα έχουν καταφέρει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κάποια σχόλια. Και να πω και δύο λόγια για την συνέχεια. Πρώτα απ' όλα, κάτι που ακούστηκε στο τελευταίο φόρουμ. Το θέμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Φάνηκε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την κοινωνία των πολιτών για το πώς λειτουργεί, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα για τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές παρεξηγήσεις, πολύ δύσκολη γραφειοκρατία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βγάλει κανείς πέρα με αυτή τη γραφειοκρατία. Για τους συμμετέχοντες, τους ζητάμε στο τέλος να μας πούνε ποιες ε, συναντήσεις ήταν πιο ενδιαφέρουσες, ποιες όχι, γιατί δεύτερη είπαν ότι ήταν πιο περίπλοκοι, πιο δύσκολοι να καταλάβουν. Οπότε νομίζω ότι για αυτά πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο. Ο ρόλος της κοινωνίας των ε, πολιτών είναι να απορροφήσει και να εκτελέσει πολλά από τα προγράμματα του ΆΜΕΤ κλπ. Και πρέπει να ξέρει κανείς πώς να το κάνει. Πολλά θέματα τέθηκαν που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας για το μέλλον. Σε πολλές χώρες δεν μπορούμε να απορροφήσουμε όλα τα χρήματα. Γιατί? Επίσης ότι όταν αλλάζει η πολιτική κατάσταση σε μια χώρα μπορεί να κόψει η κυβέρνηση, η χρηματοδότηση προγραμμάτων για τους μετανάστες. Οπότε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια ή κάποια ευελιξία ώστε η χρηματοδότηση αυτή να παραμένει. Όλα αυτά παραμένουν ανησυχία πάντα. Είναι μια μόνιμη, ένα μόνιμο θέμα. Πρέπει να βρεθούν λοιπόν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν. Τώρα για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχουμε την αρχική συζήτηση για το ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο θέμα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με την ένταξη, τη συμμετοχή, την αγορά εργασίας. Οπότε πρέπει να δούμε τώρα με τι να ασχοληθούμε αν και εσείς στη συζήτηση έχετε κάποιες ανησυχίες, να μας τι πείτε. Νομίζετε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το ένα με το άλλο θέμα, να μας το πείτε. Ευχαριστώ. Μια άλλη ιδέα είναι να δούμε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους μετανάστες, για τους πρόσφυγες. Πώς να τεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως η γενική αίσθηση είναι ότι όλοι ξέρουμε πια πολιτική κατάσταση επικρατεί. Η κοινωνία των πολιτών είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί έτσι δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα του έργου μας. Δεν καταφέρνουμε να κάνουμε τις αλλαγές. Δεν κερδίζουμε τελικά ποτέ. Οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε σε μικρές νίκες. Το επόμενο μεγάλο πράγμα που θέλουμε να πετύχουμε είναι πολλά μικρά. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά, τα πολλά μικρά. Να μιλάμε για αυτά στις κυβερνήσεις. Κάτι άλλο με το φόρουμ είναι να δούμε πώς θα πείσει τις κυβερνήσεις να ασχοληθούν περισσότερο και πώς η κοινωνία θα επικεντρωθεί περισσότερο στο τι μπορεί να κάνει ρεαλιστικές λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τόσα είπατε, λέτε δεν κερδίζουμε ποτέ, το είπατε. Σας ευχαριστώ πάντως και τις δύο για τις παρουσιάσεις σας. Θα ακούσουμε τώρα παρεμβάσεις, ερωτήσεις για οποιαδήποτε από τα μέλη του φόρουμ. Η Κριστίν Λομπονιφάη πρώτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ το Φόρουμ για τη μετανάστευση για το έργο τους. Συμφωνώ με τη φιλοσοφία των λόγων σας και με την εκθεσή σας. Η μετανάστευση δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να το δούμε σαν κάτι θετικό και λύση. Και όσο ε, καλύτερα εντάξουμε στην αγορά εργασίας του μετανίστε, τόσο το καλύτερο. Είναι πολύ βασικό αυτό για την ένταξή τους, για τη δικιά τους τη ζωή, την αξιοπρεπή, αλλά είναι σημαντικό και για οικονομικούς λόγους. Οι Ευρωπαίοι γερνούν και η δημογραφική πρόκληση είναι τεράστια. Χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο εργατικό δυναμικό. Ακούγοντάς σας, πάντως, διαπιστώνουμε ότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Κάποια πράγματα όμως έχουν ήδη ληφθεί υπόψη, τουλάχιστον εδώ. Πώς θα είναι πιο απλοποιημένη η ένταξη στην αγορά εργασίας, πώς θα μαθαίνουν οι μετανάστες στην γλώσσα της ε, χώρας, κάτι αναγκαίο για να βρουν δουλειά. Επίσης για τις συνθήκες υποδοχής έχουμε συγκίτρια την κυρία Ινχετφέλτ και ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2017 και με αυτό ζητούσαμε από τις ε, χώρες μέλη να φροντίσουν να έχουν μετανάστες με το που ζητάνε ε, άσυλο να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να δίνεται συνέχεια σε αυτό το έτομα. Οπότε, τα σχόλιά μου είναι γενικά και η ερώτησή μου. Πώς μέσα σε αυτό το δύσκολο πολιτικό κλίμα να πείσουμε ότι πρέπει να υποδεχτούμε, να βοηθήσουμε και να επενδύσουμε πάνω στους μετανάστες. Γιατί είναι η πολιτική βούληση αυτή που λείπει πάρα πολύ σήμερα. Ευχαριστώ. Να προσθέσω εδώ, Κριστίν, το θέμα είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία εδώ, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ένταξη. Είναι τόσο περίπλοκο το θέμα. Η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ένταξη είναι ήδη κάτι το περίπλοκο. Πολλοί συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Κιέγκε. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ξεκινώντας, να ευχαριστήσω. Διότι εκτίμησα ιδίω τη μνήμα που έγινε στο Global Compact, το το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Αυτό δείχνει ότι έχετε μια ε, προσέγγιση που ξεπερνά τα όρια των κρατών. Παγκόσμια. Δύο παρατηρήσεις. Όταν μιλάμε για μετανάστευση και ένταξη λοιπόν, Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και για τις νόμιμες οδούς. Για έναν απλό λόγο. Εάν θεωρούμε ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης, το σύνολό του, φέρνει μετανάστες εδώ, που αφικνούνται και παραμένουν και βρίσκονται στην επικρατεία μας χωρίς να έχουν καθεστώς πρόσφυγα, αυτό ε, απαιτεί τη λήψη κάποιων μέτρων για την ένταξή τους. Τι θα γίνει με τις νόμιμες οδούς. Η Επιτροπή μας και στην θητεία αυτή ασχολήθηκε και με μια ακόμη οδηγία για την τροποποίησή της, την γαλάζια κάρτα. Δεν είναι αρκετό, όμως είναι ένα πρώτο βήμα για να δούμε τι μπορεί να χρησιμεύσει για την κυκλοφορία, την κινητικότητα των ανθρώπων που θέλουν να έρθουν να δουλέψουν εδώ, ακόμα και αν είναι μετανάστες. Και αυτό αφορά και το στόχο του Ε, χρειάζεται πιο οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική σε επίπεδο κρατών μελών για να μπορέσουν όσοι έρχονται στην επικρατειά μας διότι μπορεί να εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους, να έχουν και εδώ κάποιο μέλλον, ε, ακόμη και εργασιακό. Βλέπω εδώ λοιπόν δύο κρίσιμα σημεία. Πρώτα απ' όλα σε επίπεδο νομικό, αλλά και ε, νομοθετικό. Όλα, το, η οικονομική κρίση έχει πλήξει τους πάντες. Ήδη είναι πολλοί οι μετανάστες στα κράτη-μέλη. Πολλοί είναι αυτοί που χάνουν τη δουλειά τους και δεν καταφέρνουν να βρουν άλλοι. Μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ξαφνικά τους ξερνάει το ίδιο το σύστημα. Πέφτουν στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος και αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευση. Θα μπορούσα να αναφέρω την περίπτωση τη Ιταλία με πολλά παραδείγματα, αλλά αυτό αφορά και άλλε χώρε. Να θυμίσω το Κάπο Βαλάτο, εκεί που πολλοί είναι αυτοί που πέφτουν θύματα τη ίδια τη αγορά εργασία διότι δεν έχουν ε, έγγραφα. Είναι λοιπόν πρόβλημα το τι γίνεται με τις χώρες που πρέπει να προσαρμοστούν, αλλά εδώ χρειάζεται και η συμμετοχή των κρατών μελών σε σχέση με τις διαδικασίες που τους ανοίγεται. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει κάπως να προσαρμόσουν τους νόμους τους, διότι διαρκώς αλλάζει γύρω μας και το τι συμβαίνει, το, το παγκόσμιο πλαίσιο και σκηνικό. Και το τελευταίο που θέλω να πω, χρειάζεται σήμερα και μια πλατφόρμα καλών πρακτικών. Πρέπει να τη συζητάμε περισσότερο, διότι υπάρχουν πάρα πολλέ καλέ πρακτικέ. Η μεγάλη πρόκληση σήμερα είναι η ένταξη. Είναι πάρα πολλέ οι καλέ πρακτικέ. Μια τεράστια πλατφόρμα γι' αυτό θα επέτρεπε το σύστημα να ε, λειτουργήσει και να εποφεληθούμε κι εμείς τα θεσμικά όργανα. Σε επίπεδο ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε, Σεσίλ. Μπάρμπαρα Σπινέλη. Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αναπτύξω και εγώ κάποια θέματα που ήδη τα άγγιξε η Σεσίλ. Καταρχάς, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Κέρια σημασία. Θα καλούσα όμως για το μέλλον να εξετάσουμε με μεγαλύτερη αυστηρότητα και κοιτάζοντας λίγο πιο σε μακρινότερους ορίζοντες το τι γίνεται με τα φαινόμενα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με την δουλεία. Εμείς καταγγέλουμε την δουλεία και τη σκλαβιά στη Λιβύη, σε άλλες χώρες, άλλες τρίτες χώρες, αλλά την έχουμε και στα πόδια μας, σπίτια μας. Το θέμα, η υπόθεση που ανέφερε η Σεσίλ του Κάπολα Ραλάτο, ας πούμε, αλλά όχι μόνο στο νότο της Ιταλίας, όλη την Ιταλική Χερσόνησο, είναι περίπτωση δουλείας, σκλαβιάς. Γνωρίζουν καλά οι συνάδελφοι τι συμβαίνει εδώ Μιλάμε για έναν τρίτο, ο οποίος ε, ως ε, μεσάζων ψάχνει δουλευ... κάποιους που θα δουλέψουν σε ένα αγρόκτημα, σε μια γεωργική εκμετάλλευση για κάποιον γεωκτήμονα. Οι λάθρομετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες πληρώνονται 15 ευρώ για μια μέρα εργασίας 15 ωρών παραβιάζοντας όλους τους κανόνες, κάτι που ταυτίζεται με την ε, δουλεία. Για να μην μιλήσουμε για την στέγαση των ε, μεταναστών αυτών στην Νότια Ιταλία, το που βρίσκονται αυτούς που τους ε, παίρνουν αυτοί οι επικεφαλής ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία «Θαύμα στο Μιλάνο» του μεταπο... της μεταπολεμικής περίοδου ε, στην Ιταλία. Εκεί όπου υπάρχει στα όρια της πόλης του Μιλάνου ένα τεράστιο αγρόκτημα με τσιφλικάδες και κολίγους. Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα από την έκθεση αυτή είναι το θέμα της ανάληψης ευθύνης από τους ίδιους τους μετανάστες, δηλαδή τι γίνεται με τις καλές πρακτικές ώστε να μπορέσουν να αυτοδιοργανωθούν στη δουλειά τους οι μετανάστες. Ιδίως ε, σε σχέση με την ε, οικονομία αλληλεγγύης και ε, είναι μια εξειδικευμένη μορφή της ε, εργασίας των μεταναστών και για τις μη κυβερνητικού οργανισμούς που αναφέρθηκαν. Υπάρχει μία που δεν αναφέρεται πολύ. Η Καθολική Εκκλησία, ιδίως στην Ιταλία. Η Καθολική Εκκλησία αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει το ρόλο του κράτους σε μεγάλο βαθμό. Το θέμα του σκάφους αυτού που βρέθηκε στην Κατάνια ε, και δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν οι μετανάστες με κυβερνητική απόφαση είναι μια υπόθεση που επιλήθηκε χάρη στην παρέμβαση της Καθολικής Εκκλησίας που ε, τελικά υποδέχτηκε τους μετανάστες και θα φροντίσει κάπου να τους εντάξει. Όμως και με την Καθολική Εκκλησία πρέπει να βρεθούν ε, κάποιο είδου συμφωνίε μεταξύ κράτους και Εκκλησίας διότι θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κρατικοί κανόνες και για τα εργασιακά δικαιώματα και τη μη διακριτική μεταχείριση ω προ τη θρησκεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Μπάρμπαρα. Δεν είναι αμφιλεγόμενο αυτό το θέμα αυτό. Όταν συζητήσαμε ε, το ζήτημα της παγκόσμιας μετανάστευσης, η Καθολική Εκκλησία είναι διαπιστωμένο γεγονός ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας ανθρωπιστικής ε, στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, οπότε δεν χρειάζεται καν να το αναφέρουμε. Η Birgit. Ευχαριστώ, Λάρα. Νομίζω ότι μπερδεύουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, η τυπική, το, το, το, το, τοπικό νομικό καθεστώς των μεταναστών που διαμένουν στις χώρες μας και το δεύτερο τι μπορούμε να κάνουμε για να τους εντάξουμε στις κοινωνίες μας και τι μπορούν να κάνουμε οι κυβερνητικές οργανώσεις για να βελτιώσουν την κατάσταση. Όσον αφορά αυτό που είπε η συνάδελφος Μπάρπαρα Σπινέλη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάσταση αυτή γιατί αφενός μιλάμε κατά κύριο λόγο και κάτι που δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν αιτούνται άσυλο, αλλά που στην πραγματικότητα το μόνο που θέλουν είναι να δουλέψουν και να βγάλουν κάποια χρήματα. Αλλά δεν έχουν το νομικό καθεστώς για να το κάνουν. Δεν έχουν επίσημη άδεια παραμονής, δεν έχουν επίσημη άδεια ε, εργασίας. Βρίσκουν όμω ανθρώπου, οι οποίοι του λένε «Ναι, έλα να δουλέψει για μένα». Και αφού δεν έχουν νομικό καθεστώς και δεν θέλουν και να ζητήσουν γιατί φοβούνται ότι θα πελαθούν, ε, γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης. Αφενό λοιπόν γίνεται μια συζήτηση σε όλα τα κράτη-μέλη μα που, που κινείται γύρω από το θέμα ότι δεν θέλουμε παράνομου μετανάστε. Από την άλλη όμω υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι Α, τι ωραία που είστε εδώ, γιατί μπορώ να σα βάλω στη δούλεψή μου υπό τι χειρότερε δυνατέ συνθήκε. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτοί και να μην λέμε ψέματα ο ένα τον άλλον. Ή θα πρέπει να πούμε στου μετανάστε που θέλουν να εργαστούν, συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε πλέον θέσει εργασία για εσά, δεν έχουμε, δεν έχουμε θέσεις εργασίας για να σα απασχολήσουμε και δυστυχώ πρέπει να σα απελάσουμε και να σα στείλουμε πίσω στι χώρε σα, ή αλλιώ να πούμε τι ωραία που είστε εδώ γιατί πράγματι υπάρχουν θέσει εργασία όπου δεν μπορούμε τις οποίες δεν μπορούμε να τις ε, καλύψουμε με υπηκόου δικού μα. Οπότε σα καλωσορίζουμε, αλλά τότε θα πρέπει να του δώσει και κανονικό, τυπικό νομικό καθεστώς για να μπορέσουν να εργαστούν υπό τι ίδιε ε, συνθήκες και τους ίδιους όρου με τους πολίτες των χωρών μας. Αυτή είναι μια γενική πολιτική απόφαση η οποία θα πρέπει να λεφθεί. Το άλλο θέμα αφορά τους ετούντε άσυλο στι χώρε μα. Εκείνοι έχουν νομικό καθεστώς και το ερώτημα είναι για ποιο λόγο δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να εργαστούν σε περίπτωση που τους χρειαζόμαστε, αν υπάρχουν δηλαδή ανοιχτές θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που ε, δεν αφορά μόνο εκείνους που έχουν ήδη το καθεστώς του ασύλου, αλλά και εκείνους που βρίσκονται σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που εξετάζονται ακόμα οι αιτήσει τους. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας, γιατί να μην τους βάλουμε να δουλέψουν. Και αυτό αφορά και τη χώρα μου. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, υπάρχουν ε, ελλείψεις ε, σε εργατικό δυναμικό εξειδικευμένο. Για ποιο λόγο να μην εκπαιδεύσουμε λοιπόν αυτού του νέου ανθρώπου που καταφθάνουν εδώ, προκειμένου να καλύψουμε αυτά τα κενά. Αυτό είναι το νομικό πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε και από εκεί και πέρα υπάρχει και η πρακτική πτυχή του θέματο για το πώ θα οργανωθούν όλα αυτά. Υπάρχουν βεβαίω και πολλέ δυσκολίε για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει να πάρουν τα κονδύλια, τον προπολογισμό, δηλαδή τα χρήματα, για να μπορέσουν να, μπορέσουν, να, μπορέσουν, με να ε, εκπαιδεύσουν ανθρώπους, να κάνουν μαθήματα γλώσσας, να οργανώσουν, να ενημερώσουν τους μετανάστες που αναζητούν δουλειά και θα πρέπει επίση να ε, εξετάσουμε και τι διαφορετικέ καταστάσει που επικρατούν στι χώρε μα. Και δεν εννοώ την πολιτική κατάσταση που πραγματικά ποικίλει και διαφέρει, αλλά τι διαφορετικέ καταστάσει για το πώ ε, είναι οργανωμένε οι χώρε μα από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο. Υπάρχει το εθνικό επίπεδο που παίρνει τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε ε, με αυτού πρέπει να μιλήσει ή, θα πρέπει, ή δίνονται τα χρήματα από το εθνικό επίπεδο στο τοπικό επίπεδο ε, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε επαφή με τις τοπικές αρχές για να μπορούμε να δούμε τι γίνονται αυτά τα χρήματα, πού καταλήγουν εν τέλει. Δεν ξέρω αν έχετε εμπειρίες εσείς συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένες όσον αφορά αυτές τις διαφορές ε, στην οργάνωση στα κράτη-μέλη και πώς αυτές οι διαφορές ενδέχεται να επηρεάζουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ή όχι. Αναφερθήκατε επίσης στο Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πράγματι και εμάς. Εξ όσων γνωρίζω όμως, υπάρχουν και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη, για την ε, χρηματοδότηση ε, δράσεων κοινωνικής ένταξης μεταναστών, όπως το Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, Συνοχής κτλ. Ε, δεν ξέρω αν έχετε τέτοια εμπειρία, να μας πείτε δηλαδή ποια ταμεία αξιοποιούνται από ποιους, ποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι τελικά να ε, επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών αν, τους, αν τις ενδιαφέρει τις διοικητικές αρχές να συνεργάζονται με μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή όχι. Ευχαριστούμε. Μπίργκετ, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να παρέμβει, θέλω και εγώ να θέσω ένα ερώτημα που αφορά την έκθεσή σας ε, την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Εγώ ε, ε έχω δουλέψει σε μη κυβερνητικέ οργανώσει, έχω υπάρξει μέλο τη Επιτροπή Απασχόληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό ε, με απασχολεί και με ανησυχεί το γεγονό ότι υπάρχει ακόμα μια τόσο έντονη πολιτική κατάσταση. υπάρχει μια πλειάδα ευρωπαϊκών ταμείων, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για παράδειγμα, το Ταμείο Συνοχής και η Κομισιόν πάντοτε μας παρακινεί, παρακινεί τα κράτη-μέλη να αξιοποιούν αυτά τα ταμεία. Υπάρχει και τώρα και το εξειδικευμένο ταμείο ε, μετανάστες και προσφύγων. Η ανησυχία μου είναι ότι βρισκόμαστε σε μια τόσο πολύ δύσκολη πολιτική κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά πρέπει να αποδειχθεί και να, και να φανεί ότι βοηθά στο θέμα της μετανάστευσης. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα έχουν εύλογη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ε, αλλά ε, πολλές φορές δεν έχουμε ακόμη καταγράψει τους μετανάστες. Μα είμαστε στο 2018 πλέον, πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι το... Δεν είμαστε στο 1987. 1988 πρέπει πλέον να, θα πρέπει κανονικά να γνωρίζουμε ποιες τοπικές αρχές, ποιες υπηρεσίες είναι υπεύθυνε για την ένταξη των ε, μεταναστών. Λέτε όμως ε, ότι πολλές φορές ε, είναι δύσκολη η χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών στα κονδύλια του Ταμείου Μετανάστευσης πόσο μάλλον στα κονδύλια των άλλων ταμείων. Ποια είναι ακριβώ συγκεκριμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Βέβαια, εντάξει, κατανοώ, πάντοτε είναι δύσκολο να έχει κανεί πρόσβαση σε κονδύλια. Προφανώ υπάρχουν κάποιοι όροι και προποθέσει για να πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μήπω θεωρείτε ότι και η δική μα επιτροπή θα έπρεπε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση. Και άλλε ε, επιτροπέ βεβαίω έχουν ερμοδιότητα και καθήκοντα γύρω από αυτά τα θέματα. Αλλά μήπω θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα σε αυτόν τον τομέα γιατί αυτά είναι σημαντικά, δεν είναι, δεν είναι απλά ε, λόγια του αέρα που θέλουμε να λέμε. Είναι πραγματικά προβλήματα στην πράξη που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας ε, στις, ε, στα κράτη-μέλη. Αφορούν ανθρώπους πραγματικούς, ακόμα και ανθρώπους δεύτερης γενιάς, όπως είναι και τα προβλήματα ρατσισμού για παράδειγμα. Επομένως θα αναρωτιόμουν μήπως μπορείτε να μας δώσετε μια καλύτερη εικόνα για το πώς ακριβώς τα κράτη-μέλη αξιοποιούν τα χρήματα, μήπως θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ίσως και η Λάουρα μπορεί να πει περισσότερο. Ξέρω βεβαίως το, το ίδιο ε, ερώτημα επαναλαμβάνεται σχεδόν από όλους πάντοτε. Τι τελικά συμβαίνει κάτω στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι που μας απασχολεί όλους. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει το λόγο. Αν κάποιο θέλει να απαντήσει, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κάντι Σούβα από την Πίκου. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτα να απαντήσω σε αυτά που ακούστηκαν εδώ για το εργατικό δυναμικό, πρόσβαση, προσδοκίες και χρηματοδότηση. Πρώτα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πιο γρήγορη, την πιο εύκολη προσδοκίες, εκμετάλλευση. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πράγματι. Η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι ότι δεν τα καταφέρνουμε. Όλα τα στοιχεία υπάρχουν, όλα τα επιχειρήματα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πούμε. Οι πολιτικές αποφάσεις όμως δεν λαμβάνονται. Παράδειγμα, είμαι Εστονή. Παρακολουθώ λοιπόν την κατάσταση στην Εστονία. Έχουμε χαμηλή μετανάστευση. Δεν έχουμε εδώ κανέναν Εστονό Ευρωβουλευτή. Υπάρχει τεράστια ανάγκη για εργατικό δυναμικό. Λείπει εργατικό δυναμικό παντού στη χώρα. Ακόμα και χαμηλών προσόντων. Υπάρχει ένα σύστημα ποσόστοσης για μετανάστες με υψηλά ε, προσόντα και το Μάρτιο είχε εξαντληθεί. Χρειάζεται δουλειά, αλλά το Μάρτιο είχε τελειώσει η ποσόστοση. Και βέβαια αρχίζουν και ακούγονται κάποιες λογικές φωνές και γράφονται διάφορα άρθρα που λένε «Μα πώς θα προχωρήσουμε, δεν έχουμε αρκετό κόσμο να δουλέψει». Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης που μπαίνουν στην ποσόστοση, αλλά υπάρχουν και άλλες θέσεις απασχόλησης για ανθρώπους χωρίς προσόντα. Για διάφορα κιόσκια, ας πούμε, λιανική πώληση, που ζητούν ξένους εργαζόμενους. Λένε δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες μας για προσωπικό χωρίς να φέρουμε ξένους. Δεν έχουμε Οπότε, τι αναγκάστηκαν να κάνουν, να ανοίγουν λιγότερες ώρες, γιατί δεν είχαν αρκετό κόσμο να καλύψει τις ώρες λειτουργίας των ε, καταστημάτων αυτών. Και αν κάποιος κάνει υπερορία, φυσικά πρέπει να πληρώνεται παραπάνω την Κυριακή στις διακοπές. Οπότε αν οι ίδιες επιχειρήσεις λένε ότι η λύση για μας είναι να έχουμε περισσότερο εργατικό δυναμικό από τη μετανάστευση. Τι έκανε όμως, ποια ήταν η απόφαση να αλλάξουν τα εργασιακά δικαιώματα. Αντί δηλαδή να λυθεί το πρόβλημα από την πλευρά της μετανάστευσης με μετανάστες, η επιλογή, η πολιτική ήταν να πάνε στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων να αλλάξει εργασιακή νομοθεσία και τώρα να είναι πιο εύκολο, να μην χρειάζεται δηλαδή να πληρώνει υπερορίες, αλλά να υπάρχει απλώς συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο για το πόσες ώρες θα δουλεύει. Άρα μπορεί να αποφασιστεί το οτιδήποτε. Αυτό αποφάσισαν οι πολιτικοί, που είναι κατά οποιασδήποτε λογική, γιατί όλοι έχουν να χάσουν από μια τέτοια ρύθμιση. Κανένα όμω πολιτικό δεν έρχεται να πει: Ωραία, να φέρουμε περισσότερου μετανάστε, αφού χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό. Όχι, γιατί οι ψηφοφόροι δεν θα συμφωνήσουν, λένε, και θα χάσουμε ψήφου. Εμεί το επιχείρημα προσπαθούμε να το πούμε και τα λέμε όλα τα επιχείρημα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η κατάσταση όμω, αδιέξοδο. Οπότε, όλοι είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία. Είναι πολύ απογοητευτικό. Τέλος πάντων, πέρα αυτό και η Λάουρα σίγουρα θα σας δώσει και άλλε πληροφορίες. Έχουν ε, γίνει και αναθεωρήσεις για το πώς θα λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζουμε να έχουμε μια καλύτερη εκδοχή τώρα. Σε ένα ιδανικό σενάριο, οι εθνικές κυβερνήσεις αποφασίζουν τον προγραμματισμό με τα χρήματα τα οποία θα παίρνουν για τις διάφορες πολιτικές που εμπίπτουν ε, στο ΑΜΙΔ. Με την κοινωνία των πολιτών, με τις τοπικές ε, κυβερνήσεις, κάτι το οποίο γίνεται σε μερικές χώρες, αλλά καθόλου σε άλλες. Οπότε, ετοιμάστε το εθνικό πρόγραμμα για το πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα, συλλογικά. Συνήθως κατευθείαν η εθνική κυβέρνηση το αποφασίζει, μερικές φορές και οι τοπικές κυβερνήσεις. Μερικές φορές οι κυβερνήσεις έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή ζητούν παράλογα πράγματα και η κοινωνία των πολιτών φτάνει να πει δεν τα θέλω αυτά τα χρήματα γιατί είναι πολύ περίπλοκο και πολύ στρεσογόνο το σύστημά σας, θα βρω χρήματα από άλλη πηγή, δεν βοηθάει τελικά. Πολύ γραφειοκρατία δηλαδή μπαίνει στο σύστημα. Και μερικές φορές οι περιορισμοί είναι τέτοιοι που είναι πάρα πολύ δύσκολο οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που συμβουλεύουν τους μετανάστες είναι δύσκολο να ξεχωρίσει το νομικό καθεστώ, γιατί δίνει συμβουλέ σε όποιον έρχεται να στη ζητήσει. Αλλά τα χρήματα αυτά κανονικά πηγαίνουν μόνο στου νόμιμου μετανάστε. Οπότε τι θα κάνει, θα ρωτήσει τον καθένα που σου έρχεται ή θα ζητήσει τα χρήματα για κάποιου πελάτε σου και όχι για κάποιου άλλου. Πώ θα δουλέψει, δηλαδή τίθενται και πρακτικά ζητήματα για τον προγραμματισμό και την σχέση με τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Κάποια χρήματα δεν απορροφώνται. Θα ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πει, μάλιστα, τα χρήματα δεν έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να δαπανηθούν, δεν θα ήταν ρελαστικό, οπότε, ωραία, αφού δεν έχουν δαπανηθεί αυτά τα χρήματα, να δούμε τι θα κάνουμε και να δει τις διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Αυτά. Η Λάουρα τώρα που είναι από την DG Home για την μετανάστευση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα. Για την χρηματοδότηση. Το έχουμε συζητήσει πράγματι πολλές φορές. Στο σημερινό ε, πλαίσιο, το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει στις χώρες μέλη. Εκείνοι δηλαδή το χρησιμοποιούν το κονδύλι, όπως γίνεται και με το κοινωνικό ταμείο και με άλλα ταμεία. Αλλά ήδη σήμερα υπάρχει μια αρχή η οποία υποχρεώνει ε, τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται στον προγραμματισμό με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με τοπικές αρχές κλπ. Ξέρουμε ότι στην πράξη αυτό λειτουργεί καλά σε κάποιες χώρες και σε κάποιες όχι δυστυχώς. Γι' αυτό και προτείνουμε να το ενισχύσουμε περισσότερο αυτό στην επόμενη πρόταση για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης προσπαθούμε να ενισχύσουμε και τη στήριξη που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές. Όχι τόσο μέσω χρηματοδότησης, αλλά ε, μπορούμε για παράδειγμα να δώσουμε μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότηση στο μέλλον. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα επανακατευθύνουμε τη χρηματοδότηση σε μερικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Δηλαδή θα δίνουμε ένα ποσό στην αρχή στις χώρες μέλη και μετά θα δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και θα υπάρχει κάποια ευελιξία. Οπότε η νέα πρόταση για το Ταμείο για την Μετανάστευση έχει διάφορες καινοτομίες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πρόσβαση στο Ταμείο, αλλά διευκρινίζει και διάφορα ζητήματα. Τώρα οι συνομοθέτες το έχουν στα χέρια τους και πιστεύω ότι θα υπάρξουν όντως βελτιώσεις. Πάντως, ήδη από σήμερα θέλω να πω ότι ένα μικρό κομμάτι του Ταμείου ε, το διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε περιοδικά κάνουμε ε, εκκλήσεις όπου συμμετέχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλοι. Υπάρχει τώρα ε, μια προσφορά για δίκτυα όπου συμμετέχουν δύο χώρες ή παραπάνω. Γιατί θέλουμε και εμείς να στηρίξουμε περισσότερο απευθείας τις τοπικές και περιφερικές αρχές και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όχι μόνο τις χώρες, τις κεντρικές αρχές. Θέλουμε λοιπόν να δουλεύουμε με διαφορετικά επίπεδα και με τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και με τις τοπικές αρχές και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τώρα πέρα από τη χρηματοδότηση, σύντομα θέλω να σας πω ότι για τις χώρες μέλη, για τη δουλειά που γίνεται, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών κτλ. Έχουμε το δίκτυο ένταξης, όπου εκεί υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για να μάθει ο ένας από τον άλλον μεταξύ των χωρών μελών. Δουλεύουμε περισσότερο με τις τοπικές ε, αρχές, στα πλαίσια των ε, αστικών στόχων του Urban Agenda. Και έχουμε εκεί και στόχους όπως είναι μια ακαδημία, έχουμε και το φόρουμ, όπου συζητάμε το θέμα της ένταξης με την κοινωνία των πολιτών. Δουλεύουμε λοιπόν σε διαφορετικά επίπεδα για την ένταξη, για να στηρίξουμε τις χώρες μέλη. Όπως είπαμε, πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα καταρχήν, αλλά κάνουμε πολλά για να στηρίξουμε και τις χώρες μέλη και τους διάφορους παράγοντες, τοπικούς, μη κυβερνητικέ ε, ε, οργανώσεις, κοινωνικούς παράγοντες, με τους ε, εργοδότες, για παράδειγμα, τους ενθαρρύνουμε να αναπτύξουν βέλτιστες πρακτικές για την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Και έχουμε και μια εταιρική σχέση με τους κοινωνικούς ε, εταίρους όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Έχουμε δηλαδή ξεκινήσει πολλές πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίξουμε το εθνικό επίπεδο, αλλά και για να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να συνεργαστούν με όλου τους παράγοντες που εμπλέκονται στο θέμα της μετανάστευσης. Ξέρω, τα πράγματα είναι πιο εύκολα αλλού, πιο δύσκολα αλλού αλλά γι' αυτό υπάρχει συνεργασία σε αυτό το δίκτυο ένταξης, προκειμένου να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να μάθουν μία από την άλλη και να εμπνευστούν από διάφορες πρακτικές και μοντέλα. Έχουμε και δραστηριότητε αμοιβαία αρρωγή στο δίκτυο αυτό, όπου οι χώρε που έχουν λιγότερη εμπειρία, η Εστονία για παράδειγμα, ζήτησε να υπάρξει μια επίσκεψη μελέτη στη Γερμανία, Πορτογαλία και άλλες χώρες ζητούν να μάθουν για το πώς γίνεται αλλού αυτή η ένταξη μεταναστών εκεί όπου πετυχαίνει. Τώρα για την νόμιμη μετανάστευση. Αυτά που είπε η και είναι ότι υπάρχει όντω ένα παράδοξο. Δηλαδή οι κυβερνήσεις παριστάνουν ότι δεν θέλουν, δεν χρειάζονται μετανάστες, ενώ στις περισσότερες χώρες μέλη λείπει εργατικό δυναμικό στις βαλτικές χώρες, ε, τις χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Αν κοιτάξετε όλα τα στοιχεία θα δείτε ότι πράγματι από τις έρευνες που γίνονται με τους, εργάτες, ε, τους, συγγνώμη, τους εργοδότες όλοι τονίζουν ότι χρειάζονται εργατικό δυναμικό. Δεν λέω ότι θα ήταν μόνο οι μετανάστες που θα κάλυπταν τις ανάγκες, υπάρχει και το εργατικό δυναμικό το τόπιο. Αλλά χρειάζεται αυτή η νόμιμη μετανάστευση για να καλύψει αυτά τα κενά. Και η Επιτροπή πάντα το έλεγε και έχουμε εμεί πρόταση για μετανάστευση υψηλών προσόντων. Υπάρχει στο τραπέζι, αλλά είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν στο Συμβούλιο χωρί μέλη. Ακόμα και αν κανεί δεν αρνείται ότι πρέπει να προσαλκύσουμε ε, μετανάστευση υψηλών προσόντων και όχι μόνο, αλλά είναι αυτό πολύ σημαντικό για την ανταγωνιστικότητά μας, την οικονομία μας, παρόλα αυτά δεν υπάρχει συμφωνία. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιχειρηματολογούμε υπέρ μιας τέτοιας απόφασης. Είμαστε και στο τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης του κεκτημένου από την νόμιμη μετανάστευση και θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα και στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή σας στους επόμενους μήνες. Οπότε έτσι ελπίζουμε να ξεκινήσει και συζήτηση για την νόμιμη μετανάστευση για να έχουμε εργατικό δυναμικό, να παραμείνει η συζήτηση ζωντανή και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο για το πώς θα αποφύγουμε τη μετανάστευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θέλετε και εσείς το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου. Στην ένταξη των μεταναστών είναι ζωτική σημασία. Συνήθω έχουμε πολύ ε, σημαντικά προγράμματα και έχουμε πολλά θέματα με τον αντίκτυπο των προγραμμάτων αυτών. Ε, επενδύουμε χρόνο, ενέργεια, αλλά σημαντικό είναι να έχουμε και ε, την κατάλληλη πρόσληψη τους μετανάστες, αν θέλουμε τα προγράμματα αυτά να είναι επιτυχημένα, τα κονδύλια μας να αποδώσουν κάτι. Γιατί εάν υπάρχει πρόθεση μάλλον να συνεργαστούμε με τι οργανώσει των μεταναστών, η απάντηση είναι ναι. <clears throat> Όμως, το θέμα είναι πώς θα λάβουν επαγγελματική ε, διάσταση οι οργανώσει των μεταναστών αυτών. Ε, για να δούμε τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των κονδυλίων αυτών και των προγραμμάτων. Συνήθω οι οργανώσει αυτέ για του μετανάστε δεν γνωρίζουν τα κονδύλια, δεν γνωρίζουν τα προγράμματα. Συνήθω οι τοπικέ αρχέ, οι τοπικοί εταίροι δεν είναι σε επαφή μαζί του. Υπάρχει έλλειψη επικοινωνία και δεν υπάρχει αρκετή συνεργασία με τι οργανώσει αυτέ. Δεύτερη παρατήρηση. Η αγορά εργασία και η ένταξη των μεταναστών εκεί όντω υπάρχει έλλειψη ε, αντιστοιχηση ε, στην αγορά εργασίας. Πολλέ είναι οι θέσεις που διατίθενται. Είναι πολύ άνεργοι, αλλά ο συνδυασμό δεν είναι καλός. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα επαγγελματικά προσόντα των μεταναστών, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας καλύτερα. Και επίσης ο ρόλος των μεταναστών επιχειρηματιών για να δημιουργηθούν για αυτούς θέσεις εργασίας 15.000 επιχειρηματίες μετανάστες είναι μέλη της οργανωσής μας. Και ξέρω ότι δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας όσο μπορούν. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει αρκετή συνεργασία με τις κοινότητες των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθούν λύσεις στα προβλήματα αυτά. Υπάρχει έλλειψη συνέστησης Υπάρχει δυσκολία να αντιληφθούν ο κόσμος πώς εργάζονται οι κοινότητες των μεταναστών. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, πολύ σημαντικό και για το μέλλον, πρέπει να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε φάση μετάβασης. Η βιομηχανική επανάσταση ξεψυχάει. Τώρα έχει αρχίσει η ψηφιακή επανάσταση. Η ψηφιακή οικονομία μπορεί να ε, δημιουργήσει περισσότερη έλευση μεταναστών ανέργων στην Ευρώπη, περισσότερο από ποτέ. Πόσο έτοιμοι είμαστε με τις πολιτικές μας, με τα εργαλεία μας, για να ετοιμάσουμε την ομάδα αυτή ανθρώπων για την αγορά εργασία του αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι για το συγκεκριμένο αυτό θέμα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ακόμη περισσότερο. αλλά νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε εδώ τον κύκλο αυτού του διαλόγου. Φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίας σας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους της ΕΜΕΤ, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη μετανάστευση. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έμειναν για τη συζήτηση του θέματος αυτού. Η ένταξη είναι ζωτική σημασία. Είναι κάτι που τώρα αρχίζει να μας αποσχολεί. Γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας φόρουμ και δεν θέλουμε να υποτιμηθεί και η δική σας παρουσία. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα. Ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Συνάδελφοι, αυτό είναι το τέλος της πρωινής συνεδρίασης. Θα σας δω την επόμενη εβδομάδα. Oh,